Good morning, colleagues. Um, we, can begin this morning with the uh, point. Καλημέρα, συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 6. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ε, σας ευχαριστώ που είστε και εδώ τελευταία μέρα πριν από τις γιορτές. Θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση της κατάστασης από τη Γενική Διεύθυνση HOME γιατί το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Στις 28 Απριλίου η Επιτροπή ενέκρινε το θεματολόγιο για την ασφάλεια, περιλαμβάνει τις βασικές δράσεις που ε, προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταπόκριση στην απάντηση στην δρομοκρατία στα πλαίσια του θεματολογίου Ευρώπη 2020. Στο θεματολόγιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι σκοπεύει να παρουσιάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πληροφορίε για την εφαρμογή του θεματολογίου. Σήμερα λοιπόν η Κομισιόν θα κάνει την πρώτη παρουσίαση για την κατάσταση τη εφαρμογή του θεματολογίου. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την κυρία Μίτση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 ε, δις ετησίως ε, για την κατάσταση της εφαρμογής. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ενημέρωση η οποία γίνεται μετά τα τραγικά γεγονότα της 13ης ε, Νοεμβρίου, γεγονότα τα οποία οδήγησαν σε επιτάχυνση κάποιων εκ των δράσεων που είχαμε στόχο να υλοποιήσουμε. Πριν περάσω στα αποτελέσματα των προηγούμενων μηνών, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το κοινό στοιχείο αυτού του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια, το οποίο τονίζει τη σχέση μεταξύ του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση των δράσεων αυτού του θεματολογίου. Και αυτό το κοινό στοιχείο είναι κάτι το οποίο έχει επισημάνει με στένος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, πιο συγκεκριμένα στο πιο πρόσφατο ψήφισμα του τον Ιούλιο φέτος. Υπάρχει επίσης ταύτιση απόψεων μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων ως προς την ουσία του θεματολογίου και επομένως ε, και ως προς τους τομείς προτεραιότητας ε, για δράσεις που θα πρέπει να μας αποσχολήσουν την επόμενη πενταετία. Και μπορώ να πω ότι αυτή η ταύτιση είναι από μόνο το ένα πρώτο επίτευγμα του θεματολογίου και μάλιστα σε ένα περιβάλλον μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ο ε, δομημένος διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Τώρα, περνάμε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Από τότε που εγκρίθηκε το θεματολόγιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Προεδρία και τα κράτη-μέλη προκειμένου να αναπτύξει ένα κοινό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της πρόοδου. Έχουμε λοιπόν ένα έγγραφο εφαρμογής, εκτέλεσης, που περιλαμβάνει τα διάφορες ομάδες ε, εργασίας του Συμβουλίου και τις επιτροπές ε, που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα για το εξάμεινο της Προεδρίας. Το έγγραφο αυτό επιτρέπει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει μια συνέπεια στις δράξεις και στους χρόνους παράδοσης και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε για να παρακολουθούμε την υπόλοιπη περίοδο ε, εφαρμογής του θεματολογίου. Να περάσουμε τώρα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια αναφέρεται στην ανάγκη να ενισχύσουμε το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα το πλαίσιο το οποίο επιτρέπει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και ε, αυξημένη συνεργασία. Γι' αυτό το 2015 συστήσαμε νέες δομές που θα μας επιτρέψουν να έχουμε ενισχυμένη και βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών και θα επιτρέψουν και ε, ανάπτυξη επιχειρησιακής συνεργασίας περαιτέρω. Έχουμε το τμήμα διαδικτύου. Στην Europol που άρχισε την πρώτη του πειραματική φάση Υπήρξε επίσης η δημιουργία του κέντρου αριστείας που άρχισε να λειτουργεί την 1η Οκτωβρίου. Το EU Internet Forum συνδυάζει εταιρείες Internet και άρχισε επίσης να λειτουργεί τον Οκτώβριο. έχει γίνει αποφασιστική πρόοδος και για τρία ακόμη σημαντικά θέματα και μητρώα για το Ευρωπαϊκό PNR και το Europol Sipol. Ως συνομοθέτης το Κοινοβούλιο έχει παίξει φυσικά αποφασιστικό ρόλο για την συμπλήρωση και ολοκλήρωση αυτών των θεμάτων. Τους περασμένους έξι μήνες επίσης θελήσαμε να διασφαλίσουμε περισσότερη συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων στον τομέα της ασφαλείας και μπορώ να σας πω ότι η ασφάλεια και οι εμπειρογνώμονες κατά της τρομοκρατίας έχουν χρησιμοποιηθεί στην αντιπροσωπή με την Τουρκία, την Ισία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και Αίγυπτο. Ε, οι διάλογοι έχουν γίνει με την Αίγυπτο, Λίβανο και Τουρκία. Πρέπει να συνεχίσουμε κύριε Πρόεδρε να σημειώνουμε περαιτέρω προόδους όπως είχαμε υποσχεθεί στο πρόγραμμα για την ασφάλεια αρχίσαμε να αναδιοργανώνουμε τις προτεραιότητες στα δημοσιονομικά μας προγράμματα για καλύτερη ευθυγράμμιση με τα, τις προτεραιότητες εσωτερικής ασφαλείας. Ο Horizon 2020 λοιπόν το πρόγραμμα του για τα έτη 16 και 17 που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο προβλέπει πολλή δουλειά για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, της βίας μάλιστα τη αυτής και αυτό έχει πραγματοποιηθεί, υλοποιηθεί με διάφορα εργαλεία σε τομείς αθλητισμού, νεολαίας κλπ. για να προωθηθούν θεμελιώδεις αξίες, η συμμετοχή των πολιτών, η ισότητα κλπ. Όσο για πρωτοβουλίες νομοθετικές της Κομισιόν, θα ήθελα να αναφέρω δύο σημαντικά θέματα. Το ένα είναι τα πυροβόλα όπλα και το άλλο η καταπολέμηση της τραμακρατίας. Για τα πυροβόλα όπλα το θέμα δεν έκρινε στις 18 Νοεμβρίου η Καμισιόν με στόχο να είναι πιο δύσκολο, δύσκολη η αγορά όπλων μέσα στην Ένωση και να υπάρχει καλύτερη χνηλασιμότης ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών, μελών και να διασφαλίζεται ότι τα όπλα που έχουν χρηστευθεί θα καταργούνται, θα παραδίδονται. Επίσης για τη λαθρεμπορία όπλων και κρυκτικών 2 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε το σχετικό κείμενο. Στις 2 Δεκεμβρίου επίσης εγκρίναμε το σχέδιο μιας νέας οδηγίας καταπολέμησης της τραμακρατίας με στόχο να γεφυρωθούν τα χάσματα που υπάρχουν και οι ελλείψεις στην νομοθεσία σχετικώς, όπως ο ορισμός της τρομοκρατικής επίθεσης καθώς και το θέμα των ξένων τρομοκρατών. E και η διασφάλιση της τιμωρίας των Τώρα η ασφάλεια των συνόρων. Εκεί καθορίστηκαν οι κοινοί δείκτες κινδύνου. Τα σύνορα θα ξανασυζητηθούν σε λίγο την Τρίτη της περασμένης εβδομάδας η Καμισιόν παρουσίασε την δέσμη μέτρων για τα σύνορα στην Ολομέλεια που θα συζητηθεί στην Λίμπε σε λίγο. Και η Επιτροπή σας θα έχει την ευκαιρία φυσικά να το συζητήσει λεπτομερώς. Και τέλος κύριε Πρόεδρέ μου, η δουλειά που κάναμε τους τελευταίους έξι μήνες είναι μόνο μια αρχή. Πολλές δραστηριότητες έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, αλλά τα αποτελέσματά τους θα φανούν τα επόμενα χρόνια. Ήδη μπορώ να σας πω ότι το 16 πολλά σημαντικά θέματα θα σας έρθουν, όπως η οδηγία για τα πυραβόλα όπλα, ή το σχέδιο οδηγία δηλαδή, καθώς και το σχέδιο οδηγία για την τραμακρατία, αλλά επίσης και για άλλους τομείς θα υποβληθούν προτάσεις. Εξών και η καταπολέμηση του δουλεμπορίου όπου το Κοινοβούλιο ανέκαθεν ναι, μας υποστήριζε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Τώρα για να μην μακρηγορήσω θα ήθελα απλώς να πω ότι τον επόμενο Μάρτιο η Καμισιόν θα υποβάλει και την πρώτη έκθεση προόδου για το θέμα αυτό του δουλεμπορίου, η λεγόμενη έκθεση Trends. Και στο τελευταίο τέταρτο του επόμενου έτους θα υποβάλουμε και έκθεση για το βαθμό στον οποίο συμμορφώνονται τα κράτη-μέλη με την οδηγία αυτή. Τέλος, έχουμε αρχίσει μια εσωτερική ανάλυση για την στρατηγική μετά το 16 ώστε να διασφαλιστεί ότι θα έχουμε καλά στοχευμένες δράσεις. Είναι αυτή η στρατηγική θα δημοσιευθεί στα τέλη του 16. Σας κατευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την προσοχή σας. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα συζητήσουμε και θα αναλύσουμε τα θέματα. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπόνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Συμφωνώ ότι οι προτεραιότητες του θεματολογίου έχουν καθοριστεί σωστά και το ερώτημα είναι πώς να εφαρμόσουμε αυτές τις προτεραιότητες ε, που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια αποτελεσματικά. Άρα, στενότερη συνεργασία ε, μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και στενότερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι περισσότερο διατεθειμένα να ανταλλάσσουν πληροφορίες, δεδομένα και να κάνουν πραγματική συνεργασία. Και εδώ θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα μια γενική ερώτηση. Τι είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο, τι σκοπεύετε να μας παραθώσετε στην αρχή του επομένου έτους, μας αναφέρατε κάποια σημεία, αλλά θα μπορούσαμε το ίσως να μας δώσετε πιο διεξοδικές πληροφορίες. Στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος, το θεματολόγιο προβλέπει την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας, ε, το οποίο υποστηρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσφατη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΑ για την ενιαψηφιακή αγορά. Τι σκοπεύετε να κάνετε ε, για το θέμα αυτό λοιπόν και αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Και η επόμενη ερώτησή μου αφορά την λειτουργία της Internet Referral Unit. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω πώς ξεκίνησε και τι σχέδια υπάρχουν για του χρόνου και αν πληρούνται όλες οι απαιτήσει. Και τέλος, σκοπεύετε να τροποποιήσετε τη βάση δεδομένων έκρης για να συμπεριλαμβάνει και δεδομένα υπηκών τρίτων χωρών. Ε, είναι αυτό μεταξύ των σχεδίων σας για το 2016 ακόμα και αν ναι, τι σκοπεύετε να κάνετε η Σοράγια Πόστ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άκουσα την Καμισιόν και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά καλά μέτρα αλλά θα ήθελα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην εσωτερική ασφάλεια, τις εσωτερικές απειλές και αναρωτιέμαι για τις απειλές μέσα στην Ένωση όπως ας πούμε η βία κατά των γενεκών Είναι πολύ σοβαρές απειλές αυτές και πολλά τα θύματα, πολλές γυναίκες και κορίτσια είναι θύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να μου πει η Καμισιόν τι σκοπεύει να κάνει για αυτή την προτεραιότητα. Μετά, τι μέτρα προβλέπονται για την ριζοσπαστικοποίηση και τους λόγους αυτής. Γιατί, γιατί υπάρχει. Για ποιον λόγο, για ποια αιτία. <coughs> παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν ανισότητες, δυσκολίες ε, στην εφαρμογή και χρήση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τι προτάσεις γίνονται για αυτό το θέμα έπειτα. Νομίζω ότι επιμένουμε υπερβολικά για τους λαθρεμπόρους και προωθητές ενώ πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα η αγορά τους να μην είναι τόσο κερδοφόρα. Τι συστάσεις θα μπορούσαν να γίνουν για να σταματήσει η δραστηριότητα αυτή χωρίς χωρίς να μπλοκά, χρειάζεται να μπλοκάρουμε την είσοδο ανθρώπων στην Ένωση. Η Σοφία Ιντεφελντ. Μάλιστα. Πάντοτε ακούω την Καμισιόν να λέει ότι κάνει νέες προτάσεις κάθε φορά που υποτίθεται ότι θα βελτιώσουν τις προϋπάρχουσες και θα κάνουν την αξιολόγηση. Αλλά δεν έχω δει πολλή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια. Ένα μέτρο μετά το άλλο, αλλά ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα τους, δεν το ξέρουμε γιατί όταν η Κομισιόν λέει ότι αξιολογεί, αξιολογεί μόνο αν μετέφεραν τις αποφάσεις καλά τα κράτη-μέλη. Δεν αξιολογούν την αποτελεσματικότητα το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα όπου ζητάει πραγματική σε βάθος αξιολόγηση των προγραμμάτων αντιμετώπισης της τρομοκρατίας πριν από τέσσερα χρόνια. Ποτέ δεν απάντησε η Καμισιόν. Το βάλαμε στο ψήφισμα και για την ε, στρατηγική της ασφάλειας φέτος. Ακόμη δεν είδα καμία απολύτως αξιολόγηση. Ξέρουμε ότι λαμβάνονται μέτρα, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το αποτέλεσμά τους. Ούτε πόσα λεφτά δίνουμε για αυτά και πόσα μας επιστρέφονται ως αποτελέσματα για την ασφάλεια. Επίσης συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία ότι η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της τραμακρατίας. Υπάρχει το θέμα της οικιακής βίας, του δουλεμπορίου ανθρώπων, του εμπορίου λευκής σαρκός κλπ. Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν αυτά που κάνουμε δεν έχουν το αντίθετο από το προσδοκόμενο αποτέλεσμα ή είναι απλώς διακοσμητικά. Ας πούμε, λέμε προώθηση των θεμελιωδών αξιών, συμφωνώ, αλλά σημειώνω επίσης ότι όλο και περισσότερες εθνικές κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα από αυτά που είπατε. Ωραία είναι όλα αυτά στα χαρτιά, αλλά δεν υπάρχουν στην πράξη. Τι κάνει λοιπόν η Καμισιόν γι' αυτό, πώς μπορεί να μας μιλάει για την προώθηση των θεμελιωδών αξιών όταν η ίδια και ο πρώτος της αντιπρόεδρος δεν είναι διατεθειμένη να μιλήσει για αυτά τα προβλήματα με τις εθνικές κυβερνήσεις. Πώς μιλάτε για προώθηση θεμελιωδών αξιών όταν ο κύριος Όρμπαν αρχίζει καμπάνια κατά των μεταναστών. Σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Πώς μπορούμε από τη μία να αγαπανούμε χρήματα και δυνατότητες για την προώθηση των θεμελιωδών αξιών ενώ ταυτόχρονα δεν αντιμετωπίζουμε τις ρίζες της άνησης μεταχείρισης και της μυσαλόδοξίας. Και αυτό είναι απειλή στην ασφάλεια, για την ασφάλειά μας. Γιατί αν υπάρχουν τέτοιες ε, διαμάχες μέσα στην κοινωνία δεν υπάρχει αρκετή ασφάλεια. Είναι λόγος άσκησης βίας. Τέλος, όταν μιλάμε για την ασφάλεια, εγώ δεν είμαι μεν δικηγόρος, αλλά όταν μιλάμε για νομοθεσία πρέπει να είναι σαφές για ποιους νομικούς όρους μιλάμε. Μιλάμε για αστυνόμευση, για δημόσια ασφάλεια, δημόσια τάξη ασφάλεια, εθνική ασφάλεια, τι ε, ζητιέται ορισμός του ναι. όρου εθνική ασφάλεια και η Κομισιόν μας λέει αυτό δεν μας νοιάζει, εθνική ασφάλεια είναι για τα κράτη-μέλη, εκείνα θα την ορίσουν. Ωραία, τότε γιατί μιλάμε για αυτά τα πράγματα ενωσιακώς. Δηλαδή, έχω ενοχληθεί γιατί η Κομισιόν συνεχώς μας κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις, ενώ δεν κάνει καμία αξιολόγηση που έχουμε ζητήσει επανειλημμένως. Ο Ντεπρέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ονοματολογία που αναφέρατε. Βέβαια δεν πρόκειται για πραγματικές προτεραιότητες, αλλά είναι τουλάχιστον μερικές λέξεις. Λοιπόν, μερικά ερωτήματα. Μιλήσατε κυρία μου για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου από τον Ιανουάριο του χρόνου. Για να λειτουργήσει αυτό το κέντρο θα έπρεπε να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Ενώ το Συμβούλιο κάλεσε την Κομισιόν να υποβάλει μία πρόταση ώστε να συνδυάζονται συστηματικά τα δεδομένα της Ευρωπόλ και της ES2. Δεν το αναφέρατε, δεν μας είπατε αν αυτή η πρόταση την επεξεργάζεστε ή αν έχει ήδη γίνει η επεξεργασία της. Και γενικότερα όλοι μας έχουμε το αίσθημα, εγώ τουλάχιστον, ότι μεγάλο τμήμα του προβλήματος με την ασφάλεια είναι ή συστηματική ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Ας πούμε Ευρωπόλ και CS2 όπως σας είπα, αλλά και το Frontex. Το Frontex δεν έχει πρόσβαση ούτε στα δεδομένα του Ευρωδάκ ούτε στους CS2. Ενώ έχουν κοινή αποστολή. Δηλαδή πρέπει και να εγγράφουν σε Μητρώα και να κατευθύνουν τους ετιτάς κάπου. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο έλλειμμα εδώ έλλειψη για τη συστηματική ανταλλαγή των πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα. Επίσης κάτι άλλο που είπατε, δύο δηλαδή, σημείωσα, αλλά αυτό είναι προσωπική μου σκέψη, τις προτάσεις σας για τα πυραβόλα όπλα. Νομίζετε σοβαρά ότι ενδυναμώνοντας για τους τίμιους πολίτες αυτή την νομοθεσία για όποιον πολίτη θέλει να αγοράσει όπλα ότι θα αντιμετωπίσετε τον εξοπλισμό των τρομοκρατών νομίζετε ότι έτσι εξοπλίζονται οι τρομοκράτες ότι οι που χρησιμοποιήθηκαν στο Παρίσι είχαν αγοραστεί από ένα απλό μαγαζί όπλων όπου πηγαίνουν οι έντιμοι πολίτε ότι κάποιος πολίτης τους τα πούλησε δηλαδή Νομίζω ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και ότι ο σοβαρότερος μηχανισμός για τον έλεγχο των όπλων θα ήταν να ενδυναμώσουμε τις ειδικευμένες υπηρεσίες που η δουλειά τους είναι να παρακολουθούν την παράνομη κυκλοφορία των όπλων αντί να παίρνετε νομοθετικά μέτρα που πλήττουν τους έντιμους πολίτας. Επίσης, αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι για την ασφάλεια στα σύνορα υπάρχει συμφωνία για τους δείκτες κοινού, κοινούς δείκτες κινδύνου οι δείκτες κοινού κινδύνου. Αυτοί οι δείκτες είναι απόρριτο ή μπορείτε να μας πείτε τίποτα παραπάνω για αυτούς. Ήδη είχα θέσει ένα σχετικό ερώτημα και άλλη φορά και η απάντηση που μου είχε δοθεί δεν ήταν πολύ ικανοποιητική. Γενικά δε, γενικά νομίζω ότι πολλές πρωτοβουλίες λαμβάνονται για την καταπολέμηση της ανασφάλειας και της τρομοκρατίας κτλ. Αλλά δεν υπάρχει πραγματική πολιτική στρατηγική δεν βλέπω να το έχετε ποτέ θέσει αυτό. Βέβαια μπορεί να μην αφορά ακριβώς εσάς το θέμα αλλά την Κομισιόν και το Συμβούλιο γενικότερα. Ευχαριστώ. Κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομη ερώτηση για την πρόταση για τα πυροβόλα όπλα και κυρίως τα ημιαυτόματα που μοιάζουν σαν αυτόματα. Πώς θα βελτιώσει η πρόταση αυτή την ασφάλειά μας. Δηλαδή να απαγορευτούν όπλα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε τρομοκρατία και σχεδόν ποτέ σε εγκλήματα. Γνωρίζετε ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν λαθρέα ε, εισαχθέντα στρατιωτικά όπλα. Μήπως πάτε να κάνετε μια ολόκληρη σταυροφορία μόνο και μόνο για να δείξετε ότι κάτι κάνετε, χωρίς να ξέρετε ακριβώς τι κάνετε. Συμφωνείτε ότι τα δικαιώματα των πολιτών μας και το δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να περιοριστεί υπερβολικά και ότι οι προτάσεις αυτές δεν προσφέρουν καμία, ε, πρόσθετη, καμία προσθέμενη αξία. κυρία Σπινέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια επιχειρήματα τα οποία έφεξε και η Σοφή και με τα οποία συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση που μας έκανε. Αλλά αντιλαμβάνομαι μεν ότι σε μερικές μέρες έχουμε Χριστούγεννα, αλλά όλη αυτή η αισιοδοξία και το να αγαπιόμαστε και αγαπάτε αλλήλους δεν με πείθει. Δεν είναι συνέντευξη τύπου αυτή εδώ, ούτε κάνουμε προπαγάνδα και αυτή η Επιτροπή, κατά την άποψή μου, πρέπει να αναφέρεται σε πράγματα χωρίς ε, να προπαγανδίζει. Και πραγματικά αυτό το οποίο θα ήθελα ε, κυρίως ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχεδόν ένα χρόνο από αυτό το θεματολόγιο για την ασφάλεια, είναι να μας πείτε τι δεν πήγε καλά. Τα αποτελέσματα δηλαδή που ζητούσε και η Σοφή δεινά. Αλλά πραγματικά θα, θα ήθελα να συζητήσουμε σοβαρά τι δεν έχει πάει καλά. Γιατί κάτι δεν πρέπει να πήγε καλά αν είχαμε τόσες τρομοκρατικές επιθέσεις. Παντού στην Ένωση υπάρχει εκμετάλλευση του φόβου από εξτρεμιστικές, εξενοφοβικές δυνάμεις οι οποίες τονίζουν στους πολίτες πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ασφάλεια, παράδειγμα χάρη. Τσεχική Δημοκρατία και Ισλαμοφοβία που την ε, προκαλεί ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ε, η Ουγγαρία, τα μέτρα τα οποία ε, ελήφθησαν ακόμα και στην Σουηδία από το Συνταγματικό Δικαστήριο που θεωρεί ότι ε, εφαρμόζει ένα καθεστώς εκτάκτου ανάγκης ε, ή τα περιστατικά βίας ε, στα hot spot κατά τη καταγραφή των μεταναστών στην Ιταλία. Και όλα αυτά τα φράγματα, όλους αυτούς τους φράχτες που διαιρούν την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι και πολύ καλά. Και πραγματικά θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά, δεν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά. Θα ήθελα να μου πείτε και τι σχέση υπάρχει μεταξύ ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και κυρίως τα θέματα της ριζοσπαστικοποίησης που σχετίζονται με το Ισλαμικό κράτος. Τι άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες από τον Ζίγμαρ Γκάμπριελ, τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας, για το ε, γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αρνείται ότι χρηματοδότησε την κατασκευή τζαμιών στην Ευρώπη. Και επίσης θα ήθελα να ξέρω και κάποια πράγματα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το ανέφερα και χθε και χθε αναφέρθηκα και στην έκθεση της Amnesty International η οποία ζητά από την Ευρώπη να αναστείλει τις συμφωνίες συνεργασίας ε, με την Τουρκία και σε θέματα ασφαλείας επειδή υπάρχει συστηματική παραβίαση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ε, διεθνών ε, συμβάσεων στην Τουρκία. Οι πρόσφυγες κατά εκατοντάδες στέλνονται σε εμπόλεμες περιοχές στη Συρία στο, και στο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ακόμα ομιλητέ στον κατάλογο. Θα κλείσω τον κατάλογο, συνάδελφοι. Η κυρία Γουίμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τις πληροφορίες που ακούσαμε. Ε, θα συμφωνήσω με την κυρία Σπινέλη ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Βλέπουμε τις διάφορες εξελίξεις Είδαμε τι έγινε, και την 11η του μηνός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει με κάποιο τρόπο ότι τα ανοιχτά σύνορα μέσα στην περιοχή Σέγγεν ενδέχεται να έχουν συμβάλει σε διευκόλυνση των επιθέσεων που σημειώθηκαν στις 13 Νοεμβρίου στο Παρίσι τελικά τι έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή τα ανοιχτά σύνορα. Ποια μέτρα προτείνει ή έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιβάλλει τις ε, αποφάσεις του Συμβουλίου. Ερώτηση, λέει ο κύριος Αγγελάρ. Ποια είναι η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Εσωτερική Στρατηγική που μάλιστα είχε εγκριθεί από το πρώτο εξάμεινο του 2010 και σύμφωνα με τις ε, διατάξεις του άρθρου 10 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τότε είδαμε πολλές εξελίξεις. Και με αυτή την εξάπλωση ενός συστήματος ανασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, να μην πω πανικό βέβαια, αλλά απέναντι στην απειλή της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας. Και επίσης και αυτή η εξάπλωση του μηνύματος μίσους της Ισλαμικής κοινότητας ή κατά της Ισλαμικής κοινότητας μέσα στην της Ισλαμικής κοινότητας μάλλον μέσα ε, και στην Ευρώπη και που χρηματοδοτείται έμεσα από την Σαουδική Αραβία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για το τελευταίο αυτό θέμα που θίξατε. Πριν επανέλθω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήθελα να επανέλθω σε αυτό το άρθρο 70 που θέτει το θέμα της έλλειψης εφαρμογής ορισμένων αποφάσεων του Συμβουλίου. Πέρα από τους εφημισμούς, η πραγματικότητα είναι ότι πολλά χρήματα πηγαίνουν στους χώρες μέλη, υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις, όμως 8 χώρες μέλη δεν ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν δεδομένα, πληροφορίες. Και αυτό που λέει ο κ. Αγγιλάρα, αλλά γνωρίζω και άλλοι συνάδελφοι, έχει σχέση και με το θέμα της παρακολούθησης του τι συμβαίνει ή με τις αποφάσεις του Συμβουλίου ε, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Ως θεματοφύλακας των συνθήκων έχει σημαντικό ρόλο να παίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προβλήματα πόρων εφόσον το Συμβούλιο δηλαδή εξακολουθεί να μην προωθεί θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και να τα χρηματοδοτεί δηλαδή. Τώρα για τα πυροβόλα όπλα για τα οποία αναφέρθηκαν ορισμένοι συνάδελφοι. Η νομική βάση έρχεται τώρα από την πλευρά της ενίας αγοράς 1-1-4 η πολιτική επιταγή έχει σχέση εδώ με την παράνομη εμπορία των όπλων. Και υπάρχει και το άρθρο 54 και στη βάση αυτού οι αρμοδιότητες μοιράζονται ανάμεσα σε δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές. Το θέμα της ενιαίας αγοράς θα ξαναπροκύψει. Για μένα ωστόσο αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα διότι προκατεί σύγχυση ανάμεσα στον στόχο των νομοθετικού στόχου δηλαδή. Βέβαια δεν είναι δικό σα θέμα τώρα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει οικοδομηθεί, ε, έχουν οικοδομηθεί τα αυτά, θα προκαλούν πρόβλημα. Ευχαριστούμε βεβαίω για την παρουσία σας εδώ και παρακαλώ να απαντήσετε στο βαθμό του δυνατού στι ερωτήσει που σας έγιναν. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής σας για τα σχόλιά τους. Νομίζω ότι με στοχοποίησαν κάπως. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα θέματα και στα σχόλια που έγιναν. Ίσως πρώτα-πρώτα για το κυβέρνο έγκλημα και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επόμενους μήνες σχετικά δηλαδή με το πώς θα εφαρμοστούν οι δράσεις που προβλέπει αυτή η προτεραιότητα. Για το 2016 προβλέπεται να γίνει πολλή δουλειά στο θέμα αυτό και σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας ο σχεδιασμός είναι να γίνει αξιολόγηση της Οδηγία του 2013 για επιθέσεις κατά των κυβερνοσυστημάτων καθώς και τις οδηγίες του 2011 για την ε, γενετήσια κατάχρηση παιδιών. Το 2016 επίσης σχεδιάζεται επανεξέταση των ε, αποφάσεων πλαισίων του 2001 για την καταπολέμηση της απάτης και την παραχάραξη ή πλαστογράφηση μέσων πληρωμής καθώς και αξιολόγηση των νομικών εμποδίων για τις ε, έρευνες, για τις ποινικές έρευνες για το κυβερνοέγκλημα με πρόσβαση σε πληροφορίες, σε αποδεικτικά στοιχεία κλπ. Προβλέπονται λοιπόν εδώ ένας αριθμός δράσεων. Μία άλλη ερώτηση ήταν σχετικά με την Internet Referral Unit της Ευρωπόλ και ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα, ας το πω που έχουμε σημειώσει τις τελευταίες εβδομάδες είχε σχέση και με την ένταξη του Interreferral Unit και των δραστηριοτήτων της μέσα στο κείμενο του κανονισμού της Ευρωπόλ. Αυτό το βήμα κρίνεται σημαντικό διότι προσφέρει ένα στέρεο νομικό πλαίσιο στην Ευρωπόλ ώστε να μπορεί να δραστηριοποιείται στον χώρο αυτό. Και ιδίω να είναι σε θέση, έχοντας προχωρήσει στην ανάλυση του υλικού και έχοντας έρθει σε επαφή με τις χώρες μέλη, να παραπέμπει το παράνομο υλικό στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και να ξεκινά αυτή η διαδικασία αφαίρεσης του παρανομιλικού από το διαδίκτυο μειώνοντας έτσι τις δυνατότητες και της ριζο, ριζοσπαστικοποίησης και της προώθησης παρόμοιων ιδεών επιγραμμικά. Σε ό,τι αφορά τώρα το σύστημα ευρωπαϊκών το, το σύστημα Equis προβλέπεται και αυτό να προχωρήσει το 2016. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιολόγηση των υφισταμένων εργαλείων, νομίζω ότι η Επιτροπή σας ήδη έχει λάβει σχετικές απαντήσεις παλαιότερα. Είναι γεγονός ότι η προηγούμενη στρατηγική εσωτερικής ασφαλείας που είχε εγκριθεί το 2010 και που κάποιος αναφέρθηκε σε αυτήν πριν από λίγο, υπήρξε αντικείμενο τριών εκθέσεων εφαρμογής το 2011, 2013 και 2014. Αυτές αξιολογούν τις δράσεις που αναλύθηκαν υπό την παλαιά εκείνη στρατηγική. Η NIN Agenda on Security βασίζεται στα συμπεράσματα εκείνων των εκθέσεων και εδώ συνδέεται και το γεγονός το οποίο αναφέρθηκαν πάλι ορισμένοι από τους βουλευτές σας στις παρεμβάσεις τους, ότι αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερη εφαρμογή, χρήση των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων. Έχουμε μηχανισμούς, εξειδικευμένους μηχανισμούς αξιολόγησης, που περιέχονται σε ορισμένα από τα νομικά μας εργαλεία, όπως οι αξιολογήσεις Schengen, που για πρώτη φορά φέτος, το 2014 δηλαδή, γίνονται από κοινού μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρών μέλων. Έχουμε και μηχανισμό αξιολογήσεως που προβλέπεται μέσα στον Ευρωπαϊκό Κύκλο Πολιτικής για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης προτίθεται να ε, καταστρώσει και δείκτες αποδοτικότητας για, την, για τον χώρο της ε, συνεργασίας στην επιβολή του δικαίου και την αντιμετώπιση των απειλών και πέραν, αυτό, πέραν αυτού μάλλον, συγγνώμη, και γι' αυτό που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε Πρόλυγου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δηλαδή ασκεί τα προνόμια που της παρέχει η συνθήκη προχωρώντας σε διαδικασίες προσφυγής αναφερθήκατε και εσείς σε μία από αυτές, στην, ε, στον χώρο της ανταλλαγής πληροφοριών. Η Κομισιόν άρχισε δηλαδή ήδη να εργάζεται πάνω σε πιλωτικά προγράμματα συνεργασίας με τις χώρες μέλη για να εξετάζει περιπτώσεις όπου η εφαρμογή φαίνεται να είναι ανεπαρκής ή ελλειπής. Άρχισε λοιπόν η Κομισιόν να το κάνει αυτό ήδη και θα συνεχιστεί το έργο αυτό του χρόνου και βεβαίως θα σας στηρούμε ενήμερους και ενήμερες. Άκουσα και ένα σχόλιο σχετικά με την Ευρωπόλ και το ΣΥΣ 2 και την διαλειτουργικότητα γενικότερα. Βέβαια αυτό είναι κέριο θέμα και πολύ σωστά το υπογραμμίσατε όταν μιλούμε για βελτίωση της ανταλλαγής προφοριών όλοι και όλες έχουμε αντιληφθεί ότι είναι σημαντικό τα εφιστάμενα συστήματα να μπορούν να συνομιλούν. Η Ευρωπόλ έχει ήδη διασύνδεση με το σύστημα SIS-2. Δίνεται τώρα ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση εάν δηλαδή η υφιστάμενη διασύνδεση και η δυνατότητα να λαμβάνονται ε, τα μηνύματα συναγερμού είναι επαρκής ή αν θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Σε ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα και όπως αναφέρεται στο κείμενο της Agenda on Security, η Κομισιόν θα παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες και τα σχέδια κυρίως μιας ομάδας χωρών μελών, σχέδιο μιας ομάδας χωρών μελών που επιτρέπουν να αυξηθεί η διαλειτουργικότητα, όχι ας το πω καλύτερα, δυνατότητα των υφισταμένων βάσεων δεδομένων επιβολής του δικαίου, του νόμου, να έχουν δηλαδή καλύτερη πρόσβαση σε παρόμοιες ή πάντως πιο ομαλή πρόσβαση και ταχύτερη σε παρόμοιες ε, βάσεις δεδομένων άλλων χωρών μελών. Αυτό βεβαίως και μέσα στα πλαίσια του Record Index. Αυτά θα τα παρακολουθούμε και τους επόμενους μήνες. Υπήρξαν ε, και αρκετές ερωτήσεις για τα πυροβόλα όπλα. Φοβάμαι ότι αυτά είναι αρκετά τεχνικά και δεν θα μπορέσω να σας δώσω μια ουσιαστική απάντηση σήμερα. Θα το αναφέρω όμως στους συναδέλφους οι οποίοι είναι ειδικοί και υπεύθυνοι για τα θέματα αυτά και βεβαίως οι προτάσεις αυτές ε, θα συζητηθούν ε, σε συγκεκριμένη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή σας και επομένως θα έρχεται και τη δυνατότητα και τότε να λάβετε καλύτερες απαντήσεις ε, στα ερωτήματά σας. Τέλος, για τους ε, δείκτες αξιολόγησης κινδύνου που αναπτύχθηκαν. Στόχος φυσικά είναι να μπορούμε να κάνουμε πιο στοχευμένους και αποτελεσματικούς ελέγχους στα σύνορα. Σαφώς και δεν είναι δεδομένα τα οποία είναι δημοσίως διαθέσιμα, ούτως ή άλλως αυτό θα ε, ε, ήταν αντίθετο στον ίδιο το σκοπό ε, ανάπτυξη αυτών των δικτών, αλλά θα το ελέγξω και αυτό, ώστε να εξετάσω σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να υπάρχει πρόσβαση για την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας κύριε Πρόεδρε. Και επίσης ε, θα ήθελα να τονίσω και κάτι τελευταίο. Δεν υπήρξε καμία πρόθεση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την παρουσίαση αυτή για προπαγάνδα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Δεν ήμουν υπερβολικά αισιόδοξη Απλώς ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ότι η κοινή συνεργασία και οι προσπάθειες ε, είναι η λύση για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Η Σοφία άλλα γρήγορα. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε είναι πολύ απογοητευτικό ως προς την εξέταση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ασφαλείας. Ε, εντάξει, είστε, έχετε καλή θέληση ως δημόσιος υπάλληλος, αλλά κατ' εμέ δεν είναι αυτή η δουλειά που πρέπει να γίνει. Πρέπει να συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο και να επιμείνουμε περισσότερο στη χορήγηση των πληροφοριών και θα ήθελα το Προεδρείο μας να υποβάλει προτάσεις στις αρχές του επόμενου έτους πώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος. Μας ζητούν να εγκρίνουμε νομοθεσία, άρα πρέπει και να εγκρίνουμε πώς η νομοθεσία αυτή θα εφαρμόζεται, αν είναι αποτελεσματική και αν εξυπηρετούμε τους πολίτες ή αν σπαταλάμε το χρόνο μας εδώ πέρα. Εδώ οι σημειώσεις μου λένε αντί να μας πληροφορεί κάποιος δημόσιος υπάλληλος να έρχεται κάποιος πολιτικά υπεύθυνος ήθελα να πω ότι χωρίς να κατηγορώ την Κομισιόν τι θέλεις Βαρβάρα ένα δευτερόλεπτο μόνο να πω ότι υποστηρίζω απόλυτα αυτό που είπε η Σοφή Ινεντβέλτ και να υπενθυμίσω απλώς ότι μόνο στη Γαλλία είχαμε 130 νεκρούς και όταν στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, έγινε μια μεγάλη επίθεση τρομοκρατική Όλη η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε για να συστήσει διερευνητικές επιτροπές, κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε και εμείς. Αν συνεχίσουμε απλώς να κάνουμε συνεδριάσεις επιτροπών που ε, ανταλλάσσουμε συγχαρητήρια, ε, νομίζω ε, ότι κάνουμε κάτι που δεν κάνουν ούτε στις ονειμένες πολιτείες που τείνουν να κρύβουν τις ευθύνες. Ευχαριστώ. Um, I'm sure that Καλά. Όχι, δεν αυτό συγχαιρόμαστε. Απλώς υπάρχουν χωριστά τμήματα της ευρωπαϊκής ε, ασφαλείας, δεν έχουν ακόμα συνδυαστεί, δεν υπάρχει συνοχή, ας πούμε τα έξυπνα σύνορα ετοιμάζονται συμβάσεις αντιτρομοκρατικές αλλά όπως είπε και ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ και η Σοφία, υπάρχει το πρόβλημα της εφαρμογής. Δεν έχουμε τις βασικές πληροφορίες από το Συμβούλιο για την ανταλλαγή πληροφοριών ας πούμε. Δεν ασχολούνται με αυτά. Σε κάθε συνεδρίασή του το Συμβούλιο δεν παίρνει αποφάσεις μπροστά στους πολίτες. Εμείς ζητήσαμε επανειλημμένως το θέμα της συνοχής. Δεν υπάρχει ακόμα συνοχή γιατί ως Επιτροπή τα συζητάμε αυτά τα πράγματα και χωρισμένος. Η νομοθεσία για τα πυραβόλα ας πούμε. Έχει δύο νομικά υπόβαθρα αυτή τη στιγμή και όχι ένα και αυτό μας δυσκολεύει και αυτό τα πράγματα. Τα μέλη λοιπόν της Επιτροπής φυσικά δεν αυτοσυγχαίρονται Προτείνω λοιπόν να είναι λίγο πιο συνολική η εξέταση. Ας πούμε, τα smart borders δεν μπορούν να εξετάζονται χωριστά από το γενικότερο θέμα της ασφαλείας. Θα ήταν λοιπόν μια πρόταση να θέσουμε στους συντονιστές την υπόθεση της οργάνωσης μιας ακρόασης στις αρχές του έτους όπου να εξετάσουμε επισταμένως το θέμα της εφαρμογής. Είναι σκανδαλώδες νομίζω ότι σοβαρές αποφάσεις δεν εφαρμόζονται και μετά να δούμε τα υπόλοιπα θέματα πτυχές της ασφαλείας. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλή πρόταση. Δεν θέλω να επιβαρύνουμε το πρόγραμμα εργασιών μας, αλλά νομίζω ότι είναι βασικό. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η Σοφή Ιντφελτ. Χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια και όχι απλώς να έρχεται κάποιος εκπρόσωπος της Κομισιόν και να θέτει τα θέματα μεμονωμένα. Αυτό ήθελα να προτείνω πριν καν να πει η Σοφία αυτά που είπε. Γιατί η εφαρμογή είναι σε πολύ άσκημη κατάσταση. Αν το δέχεστε λοιπόν συνάδελφοι, θα επανέλθουμε τον Ιανουάριο σε αυτό και θα το θέσω στους συντονιστάς. Εντάξει, εντάξει, τίποτε άλλο. Βλέπω ότι οι συντονιστές νεύουν καταφατικά. Μάλιστα. Έχουμε ήδη καθυστερήσει συνάδελφοι. Περνάμε τώρα στο 7, δηλαδή την 8η εξαμηνία έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν στο πλαίσιο της δέσμης για τα σύνορα έκανε μια έκθεση που παρατάθηκε μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου λέει για να λάβει υπόψη της τις τελευταίες εξελίξεις με τις καινούργιες ε, μεταναστευτικές ροές κλπ και τις αξιολογήσεις του Σέγγεν μεταξύ των οποίων και η τη έλεγχη. Επίσης έχει μια γνωμοδότηση για την ανάγκη αναλογικότητα στη μείωση των εσωτερικών, των εσωτερικών ελέγχων από τη Γερμανία και την Αυστρία. κύριος Ντεκόιστερ θα μας κάνει την παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι. Για το προηγούμενο σημείο ακούστηκε ότι ίσως θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο. Ίσως και για το θέμα αυτό, για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν θα πρέπει να γίνει μια πολιτική συζήτηση, αλλά φοβάμαι ότι σήμερα θα πρέπει να αρκεστείτε σε μένα. η 8η εκθέση Σέγγεν που γίνεται κάθε δύο χρόνια είναι μία από τις εκθέσεις που γίνονται από, για το λεγόμενο πακέτο δέσμη μέτρο για τα σύνορα που εγκρίθηκαν από το Σώμα των Επιτρόπων στις 5 Δεκεμβρίου. Έχουμε διάφορα στοιχεία εδώ. Υπάρχουν νομοθετικές προτάσεις, ε, καταρχάς ένας κανονισμός του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ε, ευρωπαϊκά σύνορα και την ακτοφυλακή. Υπάρχει επίσης και μία τροποποίηση στοχευμένη του άρθρου 7 της συνθήκης Σέγγεν για τους ελέγχους που θα πρέπει να γίνονται σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ε, περνούν από τα εξωτερικά σύνορα Υπάρχει επίσης και μία πολιτική ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή Συνόρων, για την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και κατόπιν υπάρχουν αρκετά άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα εκθέσεις για την κατάσταση της εφαρμογής των hot spots στην Ιταλία και στην Ελλάδα και μία έκθεση για τα Δυτικά Βαλκάνια. Όλα αυτά τα στοιχεία φυσικά είναι αλληλένδετα. Η 8 έκθεση συνήθως είναι ένας ε, έλεγχος ρουτίνας ε, της πορείας της Σέγγεν και κατά πάσα πιθανότητα θα πείτε ότι τι έλεγχος ε, της πορείας και της υγείας του Σέγγεν, ούτως ή άλλως η Σέγγεν νοσεί. Ε, θα επανέλθουμε σε αυτό στο τέλος. Συνήθως στις προηγούμενες εκθέσεις η Επιτροπή ε, ανέφερε τις πρόσφατες εξελίξεις σε όλους τους τομείς του λεγόμενου κεκτημένου Σέγγεν. Αλλά λόγω της παρούσας κατάστασης κύριε Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αλλάξει προσέγγιση. Και για παράδειγμα πρόσφατα υπήρξε συμφωνία απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων μεταξύ του Παλάου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ και με κάθε σεβασμό προς το Παλάου, αυτό δεν είναι ένα από τα στοιχεία που επηρεάζουν τη λειτουργία της θήκη Σέγγεν. Και γι' αυτό και ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της, στην έκθεσή της επικεντρώνεται σε τρία κυρίως ζητήματα λόγω του γεγονότος ότι αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο προσφυγικό ρεύμα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά και φυσικά και λόγω των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι. Υπάρχουν λοιπόν τρία ε, γενικά κεφάλαια για τη μετανάστευση και τα σύνορα και για τα εσωτερικά και για τα εξωτερικά σύνορα. Πρώτο κεφάλαιο αυτό. Δεύτερο για τις ε, τρομοκρατικές απειλές. Και ε, τελευταίο κεφάλαιο ένα κεφάλαιο το οποίο καλύπτει την εμπειρία από το πρώτο έτος λειτουργίας του νέου μηχανισμού αξιολόγησης Σέγγεν, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά, διότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα εάν τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν σωστά τα διάφορα στοιχεία τα οποία αποτελούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο που μας αφορά στο τομέα αυτό. Να ξεκινήσω λοιπόν με δύο λόγια για τη μετανάστευση και τα σύνορα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, έχουμε άνω του 1,5 εκατομμυρίου παράνομες ε, ε, εισόδους στα σύνορα ε, τον τελευταίο χρόνο. Αυτό είναι πολύ υψηλότερο από το συνολικό αριθμό των παράνομων εισόδων για το όλο διάστημα 2009-2014. Φυσικά 1,5 εκατομμύριο παράνομοι μετανάστες δεν σημαίνει, μάλλον συγγνώμη, 1,5 ε, εκατομμύριο παράνομες είσοδοι δεν σημαίνει 1,5 εκατομμύριο παράνομοι μετανάστες τμήμα των μεταναστών που ε, περιλαμβάνονται σε αυτό το 1,5 εκατομμύριο ε, έχουν μετρηθεί δύο φορές. Ε, εάν έχουν περάσει ή έχουν χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως χώρο διέλευσης και από εκεί και πέρα έχουν πάει στα, από τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ουγγαρία ή σε άλλα κράτη-μέλη, όπου εκεί και πάλι μετρήθηκαν ως παράνομοι μετανάστες. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο ήθελα να επισημάνω. Ο αριθμός αυτός ε, μας έχει οδηγήσει σε άμεση δράση, ε, για παράδειγμα με την προσέγγιση ε, και σύσταση των hot spots στην Ιταλία και στην Ελλάδα και επίσης όπως σας είπα στη δέσμη μέτρων για τα σύνορα υπάρχουν και συγκεκριμένες ειδικέ εκθέσεις για τα θέματα αυτά οι οποίες θα συζητηθούν εδώ στην Επιτροπή σας ελπίζω σύντομα. στο θεματολόγιο για τη μετανάστευση ε, περιλαμβάνονται αυτές οι δράσεις, αλλά επίσης ανακοινώθηκε ότι χρειάζεται περαιτέρω δράση προκειμένου να διαχειριστούμε καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα. Πρόκειται για έναν από τους πυλώνες ο οποίος είναι απαραίτητος ε, για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση των σύνορων. Και στη δέσμη μέτρων για τα σύνορα, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική η διαχείριση των σύνορων, υπάρχει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής ε, Σύνοριοφυλακής και ακτοφυλακής ε, και η διεύρυνση φυσικά του ε, πεδίου εφαρμογή έγκεν για το σκοπό αυτό. Ε, υποβλήθηκαν αυτά στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα, παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι θα πρέπει και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα αυτές τις προτάσεις γιατί είναι απαραίτητα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα. Κατόπιν. Έχουμε και το θέμα των εσωτερικών συνόρων, διότι οι παρανομετανάστες έχουν εισέλθει στο χώρο Σέγγεν και δεν έχουν μείνει ε, στα λεγόμενα κράτη-μέλη της πρώτης γραμμής, ε, θέλουν να περάσουν ε, στο εσωτερικό και αυτό φυσικά έχει δημιουργήσει σημαντικές δευτερεύουσες μετακινήσεις. Αυτό οδήγησε κάποια κράτη-μέλη στην ε, πανισαγωγή ελέγχων στα σύνορα, διότι αντιμετώπιζαν προβλήματα απειλές ε, για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια, λόγω του ανεξέλεγκτου αριθμού αφήξεων ε, πολλών ατόμων Πολλοί εξ αυτών ήταν ετούντες άσυλο, αλλά και μετανάστες ε, παράνομοι από τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Η Κομισιόν δημοσίευσε μια γνώμη για τη χρήση των ε, δικλείδων ασφαλείας που παρέχει το κεκτημένο Σέγγεν και θεωρεί ότι η χρήση της προσωρινής πανησαγωγή ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε αυτή την περίπτωση ήταν απαραίτητη και αναλογική. Η γνώμη πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην επανεσαγωγή ελέγχων από τη Γερμανία και την Αυστρία. Επίσης θα πρέπει να προσθέσω ότι αυτή ε, η επανεσαγωγή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν έγινε για να απαγορέσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να περάσουν τα εσωτερικά σύνορα, αλλά για να ε, διαχειριστούμε ε, με λίγο μεγαλύτερη τάξη τους ε, δευτερο, τις δευτερογενείς αυτές μετακινήσεις. Παραδείγματος χάρη, άτομα που ήθελαν να μεταβούν στη Γερμανία και να ζητήσουν άσυλο εκεί, τους κατευθύναμε προς τα σλοβενικά-αυστριακά σύνορα και μετά στα αυστριακά-γερμανικά σύνορα για να γίνουν ελέγχοι ε, υγεία, να φροντίσουμε να υπάρχουν καταβλισμοί στους οποίους θα μεταφερθούν, να τους δοθούν τρόφιμα και ρούχα και να μεταφερθούν εκεί που θέλουν να μεταφερθούν σε συνέχεια. Ε, ε, ε, Εν παρενθέσει εδώ να σας πω ότι το κεκτημένο Σέγγεν δεν είναι αυτό το οποίο δίνει δικαίωμα ε, σε έναν ετούντα να επιλέξει τη χώρα προορισμού του και εκεί που θα ζητήσει προστασία, αλλά τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν αυτό με κάποια τάξη και σειρά και έτσι υπήρχε για παράδειγμα οργανωμένη μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Τώρα υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη, πιο πρόσφατα η Σουηδία και μία από τις συνδεδεμένες χώρες, η Νορβηγία, που και αυτές επανησύγαγαν ελέγχου στα σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα σαφείς και εδώ. Οι έλεγχοι στα σύνορα, έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα δεν αποτελούν λύση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. είναι μία από τις δύο λύσεις που ε, παρέχονται στον κώδικα συνόρων Σέγγεν για να αντιμετωπίσουμε απειλές για τη δημόσια ασφάλεια και δημόσια τάξη. Αλλά ακόμα και αν όλα τα κρατημέλη επανισάγουν ελέγχους στα σύνορα, το πρόβλημα δεν θα έχει επιληθεί και ούτε και θα εξαφανιστεί. Η ροή των ετούντων άσυλο και προσφύγων θα παραμείνει, γιατί το πρόβλημα δεν το προκαλεί η Σέγγεν. Οι ρίζες του προβλήματος ε, βρίσκονται αλλού και πιο συγκεκριμένα σε κάποιες τρίτες χώρες. Η Σέγγεν λοιπόν για μας και το έχει πει σαφέστατα και ο Επίτροπός μας, δεν είναι το πρόβλημα. Η Σέγγεν όμως και κάποια τμήματα του κεκτημένου Σέγγεν θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην καλύτερη διαχείριση του προβλήματος. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα πρέπει επίσης και χωρίς να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες από αυτού, να πω ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν μια διάταξη του κώδικα σύνοραν Σέγγεν για να επανισάγουν ελέγχου στα σύνορα, προκειμένου να μπορέσουν να αναλάβουν αμέσως δράση. Υπάρχει ένα περιθώριο δύο μηνών ε, εντός ε, του οποίου ε, περιθωρίου μπορούν τα κράτη να επανεισάγουν ελέγχους. Μετά όμως η Γερμανία και η Αυστρία χρησιμοποίησαν μια άλλη διέταξη η οποία επιτρέπει επανεισαγωγή ελέγχων σε περίπτωση προβλεπόμενων γεγονότων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε ότι επειδή η κρίση διαιωνίζεται είναι αποδεκτό και μπορούν να εισάγουν ελέγχους στα σύνορα για ένα εξάμεινο ακόμα. Αυτά λοιπόν για την κατάσταση στα εσωτερικά σύνορα. Να περάσουμε τώρα στις τρομοκρατικές απειλές. Ε, αναφέρθηκε ήδη και στην προηγούμενη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε λάβει μέτρα για τους ε, κοινούς ε, δείκτες αξιολόγησης για το Ισλαμικό κράτος κλπ. Αλλά μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι, και αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό λόγω του φαινομένου των ξένων μαχητών, αποφασίστηκε να ελέγχουμε ε, τα σύνορα ε, και να ελέγχουμε άτομα και τις οικογένειές τους κατά την είσοδο και την έξοδο τους από τη χώρα. Υπάρχει λοιπόν μια συγκεκριμένη στοχευμένη πρόταση για να γίνεται αυτός ο συστηματικός έλεγχος και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και πιο αναλυτική συζήτηση όταν θα υποβληθεί η πρόταση και θα συζητηθεί στην Επιτροπή σας. Τέλος, τρίτο σκέλος της έκθεσης είναι ένας απολογισμός του πρώτου έτους εφαρμογής του νέου μηχανισμού αξιολόγησης έγκεν που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό διότι όπως σας είπα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως και σωστά ε, το υπάρχουν και εκτιμένο ώστε να συνεχίσει ο χώρος έγκεν να είναι ένας χώρος στον οποίο θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα οι άνθρωποι. Ο πρώτη διαδικασία, ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε φέτος και για να μην μακρηγορώ, οι πρώτες συστάσεις εγκρίθηκαν από το Συμβόλιο κατόπιν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και βελτιώσεις στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι συστάσεις αυτές, οι πρώτες συστάσεις εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο και έχουν διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, στις αρχές Δεκεμβρίου. Ε, που σημαίνει ότι θα μπορέσει και η Επιτροπή σας ε, να επισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τις ε, διαπιστώσεις μας στους επιτόπου ελέγχους. Εδώ τώρα θα μπορούσα να σας αναφέρω ότι πρόσφατα έγινε και μια εφηβηδιαστική επίσκεψη στην Ελλάδα, στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία αλλά και στα θαλάσσια σύνορα. Αυτή η έκθεση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και θα υποβληθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Σέγγεν προς έγκριση ε, πολύ σύντομα, διότι λόγω και της σχέσης με τα hot spots ε, και την απαραίτητη καταγραφή των μεταναστών κατά την άφηξή τους ε, μπορεί να υπάρχουν και συγκεκριμένες συνέπειες για περαιτέρω αποφάσεις ε, που θα μπορούσε να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα τη χρήση μιας συγκεκριμένη ρήτρα του κώδικα Σέγγεν που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει στο Συμβούλιο να συστήσει στα κράτη-μέλη να επανεισάγουν ελέγχους στα σύνορα προσωρινά στα εσωτερικά του σύνορα εάν υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις κατά την εφαρμογή του ε, κεκτημένου εξωτερικών συνόρων Σέγγεν. Κύριε Πρόεδρε, σας είπα ότι συνήθως εδώ κάνουμε έναν έλεγχο υγείας, ένα check-up. Και όπως σας είπα η Σέγγεν νοσεί, αλλά δεν είναι τη ασθένεια το η Σέγγεν δεν είναι το πρόβλημα, αλλά δεν είναι και η λύση. Διότι υπάρχουν και άλλοι τομεί, όπω για παράδειγμα στον τομέα πολιτική ασύλου, ε, όπου θα πρέπει να ληφθούν ε. μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόζονται πλήρω και τα υφιστάμενα μέτρα και ορθώ και ακριβώ. Ε, γι' αυτό το λόγο ότι ελπίζω στην επόμενη έκθεση της διετίας να μπορέσουμε να είμαστε λίγο πιο σαφείς ε, και να έχουμε καλύτερα ε, ε, αποτελέσματα, διότι αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να βρούμε τις λύσεις. Ευχαριστώ κύριε Σκόλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα για τη συνοπτική του παρουσίαση. Η νέα δομή της έκθεσης αυτής είναι πολύ πιο στοχευμένη από ό,τι στο παρελθόν. Πριν από έξι μήνες εδώ στην Επιτροπή μας είχα εκφράσει τη λύπη μου γιατί δεν εξετάζουμε καλύτερα τα προβλήματα αυτά. Επιτέλους έχει αρχίσει να γίνεται αυτό. Ιδιαίτερα για την κρίση των προσφύγων τους περασμένους έξι μήνες είδαμε ότι η Ένωση δεν είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τέτοια κρίση. Το πρώτο μου λοιπόν σχόλιο για τη νέα, νέο αυτό μηχανισμό αξιολόγηση του Σέντερ είναι ότι καταφέραμε από αξιολόγηση μεταξύ ισοτήμων να γίνει μια αξιολόγηση που καθοδηγείται από την Κομισιόν. Το θέμα όμως είναι τα κράτη-μέλη δεν το γνωρίζουν ή δεν θέλουν να συμμετάσχουν. Αυτό το θέτω γιατί η Κομισιόν παραδέχεται ότι 7 τουλάχιστον κράτη-μέλη δεν απανταποκρίνονται, δεν απαντούν στο ερωτηματολόγιο του Σέγγεν εγκαίρως. Ποιο δικαίωμα έχει ένα κράτος μέλος να λέει ότι υπάρχουν προβλήματα στο Σέγγεν αν δεν συνεργάζεται με το νέο μηχανισμό αξιολόγησης. Ερωτηματικό. Το έχω πει επανειλημμένος ότι Αντί να δημιουργούμε συνεχώς καινούργια εργαλεία πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα υφιστάμενα εφαρμόζονται, λειτουργούν όπως πρέπει. Άλλο θέμα για την αξιολόγηση, πρόσβαση στα αποτελέσματά της. Εντάξει, ορισμένε από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, αλλά είναι ανάγκη ολόκληρες εκθέσεις να θεωρούνται εμπιστευτικές γιατί όσο περισσότερο γνωρίζει το Κοινοβούλιο τι συμβαίνει, τόσο καλύτερα θα ξεωρίζει τι μέτρα χρειάζονται. Η έκθεση ήδη δείχνει ότι τα πρώτα αποτελέσματα του νέου μηχανισμού αξιολόγηση με, τις σχεδιαζόμενες, με τους προβλεπόμενους ελέγχους. Υπάρχουν μερικές βελτιώσεις βέβαια που μπορούν να γίνουν ιδίως για το CS2 που παραδέχεται η Κομισιόν ότι δεν χρησιμοποιείται επαρκώς. Επίσης, δέχομαι την ιδέα των τον ελέγχων στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στα σύνορα με την Ουγγαρία και όλους τις τους γείτονες, αλλά τώρα και στα γαλλογερμανικά. Τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα όμως δεν είναι προφανή. Μπορεί να μας πει η Κομισιόν πότε θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι και αν θα είναι ισοδύναμοι με ελέγχους στα σύνορα. Έχετε καμία πληροφόρηση. Αυτά τα θέματα συνδέονται με την επανάληψη, την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων σε διάφορες χώρες. Αυτό οφείλεται βέβαια στην κρίση των προσφύγων, αλλά έχω συγκεκριμένα ερωτήματα. Φαίνεται ότι μόνο η Σλοβενία υπέβαλε εκθέσεις για τα αποτελέσματα της επαναφοράς των ελέγχων της όπως απαιτεί το άρθρο 29 του Σέγγεν. Η Καμισιόν γνωρίζει πότε θα λάβουμε ανάλογες εκθέσεις από άλλες χώρες μέλη. Εκτός αυτού πιστεύει ότι υπήρξε επαρκή σύνδεση και συνεννόηση μεταξύ των χωρών μελών για αυτό το θέμα των συνοριακών ελέγχων. Γιατί φαίνεται ότι ο ένας ακολουθούσε τον άλλον. Είναι φανερό ότι μερικές χώρες επανέφεραν τους ελέγχους για να διαχειριστούν καλύτερα τις μεταναστευτικές ροές, άλλες όμως απλώς για να κλείσουν τα σύνορά τους. Θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι η Καμισιόν θεωρεί ότι η επαναφορά των ελέγχων δεν παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, αλλά πρέπει να είναι δε δικαιολογημένη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως καθώς όλο και περισσότερες μικρές χώρες ανακοινώνουν παρόμοια μέτρα. Είναι προφανές για όλους ότι το Σέγγεν πιέζεται, αλλά πρέπει να έχουμε μια σαφή και αληθινή εικόνα της πραγματικότητας. Πρέπει η Κομισιόν να, υπάρχουν αντιδράσει στεναρά, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει για την εκμετάλλευση και εκτιμένη του Σέγγεν στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ξεκάθαρη αυτή ανάπτυξη του θέματος και ενημέρωση. Όλοι έχουμε σημαντικές ανησυχίες και εσείς αναγνωρίζετε ότι νοσεί το σύστημα Σέγγεν σήμερα. Όλα σχεδόν τα μέτρα, όλα τα hot spot, οι επιστροφές και τα αυτά δεν αποδίδουν. Ναι. Ξέρετε ότι είμαι από τη Σλοβενία. Είμαι Σλοβένα Ευρωβουλευτή και μόλις μιλήσατε για, τις, για τους φράχτες. Είναι οδυνηρό για μας. Έχουμε φτιάξει πράγματι φράχτε από αγκαθωτά σηματοπλέγματα στα σύνορά μας και η κοινωνία μας είναι πολύ διχασμένη. Νιώθουμε από την αρχή ότι αναγκαστήκαμε να φτιάξουμε τους φράχτες γιατί δεν ήταν επαρκή τα μέτρα. Ως μικρή χώρα δεν καταρθώσαμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα ρεύματα των ανθρώπων που έρχονταν τώρα βέβαια, χειμώνα, ο κόσμος που έρχεται λιγότερο. την άνοιξη αναμένουμε νέα κύματα, κυρίω από την οδό των Βαλκανίων. Εάν τα μέτρα δεν αποδειχθούν επαρκή, αυτό που βλέπουμε ωστόσο είναι καθημερινές διαδηλώσει στα σύνορα. Ε, εμείς ε, χάνουμε και οικονομικά και συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών. Σε όλα αυτά τα μέτωπα χάνουμε. Και υπάρχει και ένας αυξανόμενος φόβος τι θα γίνει με την συνθήκη Σέγγεν. Από τη στιγμή που αρχίσουν να ανοιγείρονται φράχτες στα σύνορα, είναι καθαρό ότι θα είναι δύσκολο να αφαιρεθούν. Πότε θα αφαιρεθούν οι φράχτες, δηλαδή πώς, τι θα προκαλέσει την αφαίρεσή τους. Έχουμε όλο και περισσότερους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Η ερώτησή μου είναι, γνωρίζω τη θέση σας βέβαια και είπε και ο Παύλο Κοέλιο σχετικά για τους φράχτες στην Ευρώπη. Όμω πόσο σοβαρές είναι οι ανησυχίες ότι κινούμεθα προς ένα μίνι Σέγγεν. Νομικά είναι δυνατόν αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι που ε, πρέπει να το απορρίψουμε με κάθε τρόπο, διότι θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ωστόσο οι ανησυχίες υπάρχουν. Έχω τώρα ορισμένε συγκεκριμένε ερωτήσεις. Είναι σαφές για μένα ότι οι φράχτες δεν λύνουν το πρόβλημα. Όταν άρχισε η Ουγγαρία να ορθώνει φράχτες, το μόνο που κατάφεραν ήταν να στρέψουν τα ρεύματα προς άλλες χώρες. Αυτό συμβαίνει. Η Ευρώπη είναι χώρα προς την οποία θα κατευθύνονται τα μεταναστευτικά ρεύματα και θα έρχονται οι άνθρωποι. Εγώ δεν βλέπω ε, μέλλον της Ευρώπης με φράχτες. Όταν είδαμε τις πρώτες 100-200 ανθρώπους να έρχονται στη Σλοβενία δεν υπήρχε καταγραφή ούτε ε, συλλογή των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πώς θα επανέλθουμε λοιπόν στο καθεστώς αυτό. Ακόμη και πρόσφατα που μίλησα με εκπροσώπους των σερβικών αρχών αυτοί παίρνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Όμως δεν συνδέονται με το σύστημα Ευρωντάκ και τα υπόλοιπα γιατί το κάνουν τότε. Πώς θα λυθούν αυτά τα πρακτικά θέματα. Αυτοί ό,τι καταγραφή και να κάνουν, τα δεδομένα μένουν εκεί, στη χώρα τους. Ίσως λοιπόν μπορείτε να με βοηθήσετε να απαντήσω στο ερώτημα αυτό, γιατί εγώ δεν έχω ξεκάθαρη απάντηση. Μετά οι ανθρωπιστικές βίζες, τα είπε κάποιος πριν. Αναθεώρηση του κώδικα προξενικών θεωρήσεων. Είπαμε να μπουν εκεί και πράγματα για τις ανθρωπιστικές βίζες. Μπορεί να σωθούν χιλιάδες ζωές αντί οι άνθρωποι να προσπαθούν να διέλθουν από τη Μεσόγειο να παίρνουν ανθρωπιστικές βίζες. Γιατί δεν είναι υπέρ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζω βέβαια λίγο πολύ την απάντηση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ασκήσω κάποια πίεση για το θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Γιατί υπάρχουν, ε, είναι σωστό να υπάρχουν κάποιες νόμιμες διαδρομές προς την Ευρώπη. Ποιες θα είναι τώρα οι επιπτώσεις της ε, εφαρμογής των αποφάσεων ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αναγκαστική επιστροφή, compulsory, compulsory reallocation, μετεγκατάσταση μάλλον, για ορισμένε χώρες όπως η δική μου, θα δούμε ότι οι περισσότερες χώρες μέλη δεν δρούν, αντιδρούν. Και γι' αυτό καταραίει το σύστημα Schengen. Τώρα, υπάρχει προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την μετεγκατάσταση. Ποια θα είναι η επίπτωση της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν θα συνεχίσω παρόλο που και άλλε ερωτήσεις για να δώσω το, λόγο και σε, το χρόνο και σε άλλου. Κοράτσα Εγώ ανησυχώ πολύ για την κατάσταση τη ε, συνθήκης Σέγγεν και γι' αυτό με ικανοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση αυτή με πολύ προσεκτικό τρόπο και είναι ανοιχτή απέναντί μας. Για να εφαρμοστεί ο κώδικας Σέγγεν δεν πρέπει να κλείσουν τα σύνορα, ούτε να γύρονται φράχτες. Το γεγονός ότι οι χώρες μέρη μπορούν να κάνουν και κατάχρηση των δυνατότητων αυτών, αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος. Δεν βελτιώνει τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ούτε καταπολεμείται η τρομοκρατία έτσι. Η ελευθερία διακινήσεως του Σέγγεν, μέσα στο χώρο Σέγγεν δηλαδή, είναι από τα μεγαλύτερά μας επιτεύγματα. Θα πρέπει με κοινή προσπάθεια υπερκομματική και υπερεθνική να επιμείνουμε, να διατηρηθούν αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται σεβασμός του κώδικα Σέγγεν, χρειάζεται ενίσχυσή του και γι' αυτό χαίρομαι για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση του κώδικα Σέγγεν Ελέγχου ε, εισοδου εισόδου-εξόδου και για Ευρωπαίου πολίτε. και να επανέλθουμε σε αυτό που είπατε εσεί κύριε Πρόεδρε, δηλαδή εφαρμογή. Να πω στην Κριστίνα ότι δεν είναι η Ευρώπη εκείνη η οποία δεν πάει καλά. Οι χώρες μέλη δεν πάνε καλά. Ο εθνικισμός είναι το πρόβλημα. Ο προστατευτισμός είναι το πρόβλημα. Όχι η ίδια η Ευρώπη διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τη δουλειά της. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας παρά τις πολιτικές αντιθέσεις μας και μπορώ να σας πω και άλλα πράγματα για αυτές, αλλά οι κυβερνήσεις δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις. Εάν έχετε κοινέ νομοθετικές διατάξεις, συμφωνίες, εφόσον έχετε το Συμβούλιο που λαμβάνει μια κοινή απόφαση και μετά οι μισές χώρες μέλη δεν τις εφαρμόζουν, ε τότε που φταίει η Ευρώπη. Γιατί έχουμε αυτή την κατάσταση του Σέγγεν, κύριε Πρόεδρε, πληρώνουμε ένα τίμημα προσπαθούμε να βουλώσουμε τις τρύπες που αφήνουν οι χώρες μέλη μην λαμβάνοντας ε, υπόψη τις ευθύνης τους. Είναι σαν το ευρώ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η ζώνη ευρώ εάν οι χώρες μέλη δεν προβαίνουν σε μεταρρυθμίσεις και βλέπουμε τι γίνεται. Εάν τώρα θεωρήσετε ότι λειτουργεί το σύστημα Schengen αλλά είναι εντελώς ανοιχτά τα εξωτερικά σύνορα, ε, πώς θα γίνει. Όταν εμείς πηγαίνουμε σε τρίτες χώρες, μας ζητούν τα ταξιδιωτικά μας έγγραφα. Γιατί να έρχονται από αλλού άνθρωποι χωρίς καμία καταγραφή, χωρίς κανέναν έλεγχο. Τα συζητήσαμε αυτά και την προηγούμενη εβδομάδα. Χρειάζεται ενίσχυση του Frontex. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ στην Ευρώπη πρέπει να καταγράφονται, να ταυτοποιούνται, να λαμβάνονται τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Και όλα τα έγγραφα, βιομετρικά, διαβατήρια κλπ. πρέπει να καταχωρίζονται. Όχι απλώς να τα κοιτούν οι ελεγκτές, μια να μια ματιά, αυτή είναι η προπόθεση για να λειτουργήσει η Σέγγεν. Έρχομαι τώρα σε αυτά που είπε η κυρία Σπινέλη πριν για την κατάσταση στην Σουηδία, γιατί δεν έλαβα το λόγο στην προηγούμενη συζήτηση. Δεν είναι το συνταγματικό δικαστήριο εκείνο το οποίο απεφάνθη, δεν είναι δικαστικό όργανο. Το Log στο σουηδικό σύστημα έχει ως εξής. Σε κάθε προτινόμενη νομοθεσία υπάρχει ένα νομικό όργανο, το οποίο όμως δεν είναι δικαστικό, είναι οργανισμός της κυβερνήσεως που εξετάζει το νομοσχέδιο και αποφαίνεται. Και λέει λοιπόν ότι αυτά τα νέα μέτρα είναι νέα δέσμη, απελπισμένη, απελπισμένη νέα δέσμη μέτρων της κυβερνήσεως, ότι είναι υπερβολική, για μέτρα δηλαδή στα σύνορα. Εγώ δεν υποστηρίζω την θέση της κυβερνήσεως. Εγώ νομίζω όμως ότι εδώ πρέπει να λεχθούν δύο πράγματα. Η Σουηδία υπήρξε η πιο γενναιόδορη χώρα στην Ευρώπη τα τελευταία 3-4 χρόνια. Φέτος δέχεται πάνω από 160.000 ετούντες άσυλο. Από αυτούς πάνω από 32.000 είναι ασυνόδευτα παιδιά. Στη διάρκεια του Νοεμβρίου πάνω από 10.000 ερχόντουσαν κάθε εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό. Η Σουηδία αντιμετωπίζει την πρόκληση να είναι η πρώτη χώρα Άφηξη. Γιατί, διότι οι άλλες με μέσα από τις οποίες διήλθαν αυτοί δεν τους καταγράφουν και επομένω αντιμετωπίζει η Σουηδία την πρόκληση να είναι ταυτόχρονα και η τελική χώρα προορισμού, δηλαδή ένταξη στην αγορά εργασίας και όλα τα σχετικά. Δέχεται λοιπόν τι ανάλογε πιέσει η Σουηδία. Η χώρες μέλη αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αγνοήσει το γεγονός ότι η Σουηδία και αυτή χρειάζεται βοήθεια. Και να τα αποτελέσματα. Έχουμε τώρα απόφαση από την κυβέρνηση, μάλιστα πράσινη κυβέρνηση, πράσινη και κόκκινη είναι αυτή η κυβέρνηση, έτσι, προσέξτε, που στην ουσία κάνει αυτά που προτείνει η άκρα δεξιά. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι άσχημο. Ρωτώ λοιπόν, παρακαλώ μάλλον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εξετάσει πολύ προσεκτικά την απόφαση που έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα η Σουηδική κυβέρνηση να επαναφέρει συνοριακούς ελέγχους έλεγχο στην γέφυρα Όρεσουγκ για κάθε είδους ε, δημόσιο μεταφορικό μέσο, λεωφορεία, τρένα και Η απόφαση αυτή λήφθηκε για μια τριετία και είναι νόμος. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορείτε παρακαλώ να εξετάσετε εάν αυτό παραβαίνει τη συνθήκη του Σένγεν. Είπατε πριν από λίγο ότι τα μέγιστα όρια είναι, τα ανώτατα όρια είναι 2 ή 6 μηνών. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μια έκτακτη δυνατότητα που επιτρέπει 2 χρόνια. Όμως χρειάζεται μια διευκρίνηση και χρειάζεται αυτή η στάτη καταφυγή που είναι το κριτήριο της δημόσιας ασφάλειας να γίνεται σεβαστό. Αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν έκανε την παρουσίασή τη η Κομισιόν, είδα τα μηνύματά μου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γιατί κάθε μια-δυο μέρε παίρνουμε επιστολέ για κράτη-μέλη που έχουν ξεκινήσει ελέγχου συνόρων. Και εγώ μέτρησα 8 κράτη-μέλη. Μάλτα, Νορβηγία, Σλοβενία, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία και Ουγγαρία. Και μετά ο Κάρλο Κοέγιο αναφέρθηκε το ενδεχόμενο και η χώρα μου, οι κάτω χώρες να κάνουν ελέγχου στα γερμανικά σύνορα. Ναι, κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, έχω δει και κάποιες περιπτώσεις τις οποίες ε, το είπαν και στο ραδιόφωνο. Περνούν τα σύνορα, φτάνουν στο Βέλγιο, παρκάρουν ε, σε ένα χώρο στάθμευσης ε, δίπλα στο δρόμο και μετά μέσω ασυρμάτου λένε στους φίλους τους στα Ολλανδικά σύνορα περνάει ένα αυτοκίνητο, ε, βλέπω ότι η πινακίδα είναι από χώρα της Ανατολικής Ευρώπης και το σταματάνε και λένε ότι το κάνουν από ένστικτο. Ναι. Ε, επομένως υπάρχουν συνοριοφύλακες οι οποίοι πηγαίνουν στο Βέλγιο και εργάζονται ε, και ενημερώνουν τις κάτω χώρες και επιλέγουν βάσει ενστίκτου. Πραγματικά εγώ έχω πρόβλημα, έθεσα σχετική ερώτηση στην Ολλανδική κυβέρνηση και είπαν ότι όλα είναι ε, στα πλαίσια του νόμου. Δεν νομίζω ότι το να επιλέγουμε βάση ενστίκτου ε, είναι βάση νόμου. Νομίζω το πρόβλημα δεν είναι αν και οι οκτώ χώρες και η χώρα μου λειτουργούν βάση νόμου, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ε, χάνεται η κατανόηση και ο ενθουσιασμός για τη Σέγγεν. Πριν από κανένα δυο εβδομάδες οι εφημερίδες έλεγαν ότι τα κράτη-μέλη θα πάνε στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και έλεγαν ότι η Ελλάδα προσωρινά θα διωχθεί από τη Σέγγεν. Δεν συνέβη τίποτα, αλλά είχαν γεμίσει εφημερίδες και αυτή είναι και ε, λανθασμένη χρήση της έκφρασης που θα χρησιμοποιήσω κύριε Πρόεδρε. Το έγραφαν όλες οι εφημερίδες και το θέμα είναι ότι επειδή ακριβώ το έγραψαν, το κακό έγινε. Το Κοινοβούλιο είναι υπέρ της Σέγγεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μάχη για τη Σέγγεν, αλλά το θέμα είναι ότι ο εταίρος που δεν είναι εδώ σήμερα, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη, φαίνεται να μην απασχολείται καθόλου για το γεγονός ότι ζημιώνεται η κατάσταση και ε, η, τα όσα γράφονται στον τύπο ουσιαστικά οδηγούν σε λιγότερη υποστήριξη για τη Σέγγεν. Και νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά που μας αναλογεί για το μέλλον. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το σκεπτικό, πώς μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να σταματήσουν να ε, κάνουν προτάσεις ε, αυτής του είδου και να σταματήσουν ε, και τους ελέγχους. Πρόκειται για 8 χώρες. Η Μάλτα γιατί έχει επανεισάγει ελέγχους. Ε, πού είναι τα εσωτερικά της σύνορα. Γύρω-γύρω νερά έχει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντεκοστέρ, εσείς προβλέψατε ότι ε, θα πρέπει να γίνει πολιτική συζήτηση και αυτό κάνω κι εγώ. Είμαστε εδώ για να κάνουμε δηλώσεις και θα ήθελα να σας ζητήσω να το διαβιβάσετε στους υψηλά πολιτικούς συσταμένους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι εμείς εκπροσωπούμε εδώ τους Ευρωπαίους πολίτες που ανησυχούν για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κεκτημένο Σέγγεν, που θεωρείται το πολυτιμότερο αγαθό της ευρωπαϊκής εμπειρίας μέχρι τούδε. Σύμφωνα με τις φυγμομετρήσεις δεν υπάρχει τίποτα άλλο το οποίο να αγαπούν περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες από το κοινοτικό κεκτημένο. Και το είπατε, η Σέγγεν νοσεί, πεθαίνει, θα τη γλιτώσει, ε, χάνεται σιγά σιγά, θα εξαφανιστεί χωρίς ε, να ρωτήσει τα, από τα κράτη -μέλη, να ζητήσει συγγνώμη από τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να φροντίσουν οποιαδήποτε αναστολή στη Σέγγεν ε, να είναι προσωρινή. και αυτή η επαναφορά των εσωτερικών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πράγματι προσωρινή. Είμαστε έτοιμοι να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασώσουμε το κεκτημένο Σέγγεν. Διότι η άποψη πολλών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι η Σέγγεν χάνεται σιγά σιγά. Ότι επαναφέρουμε τους ελέγχους στα σύνορα, ελέγχους ταυτότητας, ε, εξακρίβωση στοιχείων σε κάθε ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, ακόμα και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Το θέμα είναι πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε διαδικασία επί παραβάση και οποιοδήποτε έλεγχο ώστε να δράσει ως πραγματικός θεματοφύλακας των συνθήκων ώστε τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν να τηρήσουν μόνο αυτό το προσωρινό ε, στοιχείο και να μπορούμε να πούμε λοιπόν ε, στους πολίτες ότι είναι ε, προσωρινό και δεν θα μονιμοποιηθεί διότι ουδέν μονιμότερο το προσωρινό. Ε, ώστε να είναι βέβαιοι ότι αυτά τα προσωρινά μέτρα put down δεν θα παραταθούν ώστε ε, να αντιμετωπίσουμε και εμείς ε, τους ε, ελέγχους ασφαλείας και να μην μονιμοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Αυτό είναι το μήνυμα λοιπόν το οποίο θα ήθελα να μεταφέρετε στους υψηλά εσταμένους ανωτέρους σας. Ευχαριστώ κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Δεκέστερ είναι εγνωσμένο κύριο υπάλληλο, αλλά νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον τμήμα της παρέμβασής του ήταν όταν μας είπε στην αρχή ότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα θα έπρεπε να γίνει σε πολιτικό επίπεδο, διότι αυτή είναι η ουσία. Η Σέγγεν είναι πολιτικό πρόβλημα, δεν είναι μόνο διοικητικό θέμα. Νομίζω ότι είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Εγώ είμαι υπέρμαχος ε, ασυζητητή της Σέγγεν. Πιστεύω ότι η Σέγγεν ε, βουλιάζει, η Ευρώπη θα διαλυθεί και θα διαλυθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η απόλυτη πεποίθησή μου. Η Σέγγεν έχει δύο στοιχεία, τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και την ελευθερή κυκλοφορία. Ελάτε στη θέση ενό πολίτη που του λέμε «Ξέρετε, υπάρχει ένα κοινό εξωτερικό σύνορο και το ελέγχουμε». Και ταυτόχρονα μαθαίνει ότι υπάρχουν και 1,5 εκατομμύριο παράνομοι μετανάστες. Πώς θα πιστέψει ότι υπάρχουν ένα κοινό σύνορο που ελέγχεται με 1,5 εκατομμύριο παράνομους μετανάστες που μπήκαν σε ένα χρόνο. Και από την άλλη μεριά του λέμε ότι προσπαθούμε να διασώσουμε την ε, εσωτερική ασφάλεια και κάθε μέρα ακούν ότι η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ελβετία επαναφέρουν του ελέγχου στα σύνορα και μάλιστα βλέπουν και εικόνες όπου ε, έχουν βάλει και ε, σειρματοπλέγματα οι χώρες ε, στα σύνορα. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε τι σημαίνει αυτό για τη συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών, το να βλέπουν σειρματοπλέγματα η απάντηση δεν μπορεί να είναι απλώς γραφειοκρατική, πρέπει να είναι πολιτική. Να σας αναφέρω δύο περιπτώσεις. Την περίπτωση των ελέγχων των εξωτερικών συνόρων, ε, Είχαμε δύο ελέγχου, 8-9, δεν ξέρω αν δουλεύουν αποτελεσματικά, αν κάνουν δουλειά τους σωστά και ποιος είναι ο στόχος. Έχω και ένα ακόμα ε, παράδειγμα, αυτά στο Notepad Calais που δεν λειτουργεί τίποτα. Υπάρχει και κάτι άλλο. Οι Καναδοί υποδέχθηκαν 25.000 υποψήφιους πολιτικούς πρόσφυγες. Και τι έκαναν, μία εναέρια γέφυρα. Πήγαν, τους πήραν και τους έφεραν με αεροπλάνο στον Καναδά. Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο. Για, ε, δεν είναι απαραίτητα ε, με αεροπλάνο γιατί είμαστε πολύ κοντά. Αλλά ε, θα έρχονται ατάκτως εάν δεν κάνουμε κάτι για να προβλέψουμε την άφηξή τους. Ε, τα εξωτερικά σύνορα λοιπόν μετά δεν θα είναι απλώς ανεξέλεγκτα. Θα πιστεύει ο κόσμος ότι μπορεί να μπει ο πάσα ένας για να μην πω και χειρότερα. Επομένως, να υπάρχει ένας νόμιμος τρόπος να μπουν στο χώρο σε οι πρόσφυγες. Αυτό είναι απαραίτητο. Δεν ξέρω αν θα είναι ανθρωπιστική βίζα ή οποιοδήποτε άλλο. Ε, κύριε Ντεκοστέρ, να σας πω ότι η ανθρωπιστική βίζα δεν θα πρέπει να βρίσκεται στον Κοντέγγεν, ε, ναι, έτσι μας είπατε, αλλά αν δεν είναι εκεί, πού θα πρέπει να είναι. Έχετε κάποια πρόταση. Αν έχετε πρόταση, να μας την κάνετε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλα μέσα στη διάθεσή μας και επομένως προτείνω ότι θα πρέπει να δοθεί μια σοβαρή μάχη, ώστε να υπάρχει μια νόμιμη οδός εισόδου των προσφύγων. Ε, διότι πρόκειται για κάτι το οποίο θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια και θα αποσταθεροποιήσει σε πολιτικό επίπεδο τις χώρες μας. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στο πολιτικό επίπεδο. Α, θα σταθώ σε ένα στοιχείο ασφαλείας εδώ. Είπαμε ότι θα επαναφέρουμε του ελέγχου στα σύνορα. Οι Γάλλοι είχαν έλεγχο στα σύνορα την ημέρα που μπήκαν οι τρομοκράτε από το Βέλγιο για την επίθεση και δεν του σταμάτησαν γιατί, γιατί δεν είχαν τις σωστέ πληροφορίε. Τώρα θα επαναφέρουμε τους συστηματικούς ελέγχους των Ευρωπαίων στα εξωτερικά σύνολα. Ευρωπαίων, έτσι, το οποίο νομίζω ότι φύγει και την ελεύθερη κυκλοφορία. Για λόγους ασφαλείας, θεωρητικά για να εντοπίσουμε τους ε, ε, τρομοκράτες. Πώς θα τους βρούμε αυτούς. Πρέπει να ψάξουμε στις δα Τους σοσιαλιστές, λέει ο μιλητής. Τι είπα. Να εντοπίσουμε ποιους Ακούσαμε τους σοσιαλιστές. Δεν είπα τους σοσιαλιστές, είπα. Ε, συγγνώμη, συγγνώμη. Τους τρομοκράτες, ε, δεν ήθελα να πω τους σοσιαλιστές. Ε, συγγνώμη, ποτέ δεν θα συσχέτιζα σοσιαλιστές με τρομοκράτες. Συγγνώμη, σας έκοψα την ανάσα, αλλά μπορείτε να ξαναναπνέσετε Συγγνώμη. Τέλος πάντων, χάθηκε και το επιχείρημα. Λοιπόν, θα ελέγχουμε όλου του Ευρωπαίου πολίτε, αλλά για να δούμε αν είναι τρομοκράτε, το είπα καλά τώρα. Για να δούμε αν είναι τρομοκράτε, θα πρέπει να ελέγξουμε τι πληροφορίε στιγμή που περνούν με βάση δεδομένων. Το ΣΥΣ. Τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν ε, εισάγει όλε τι απαραίτητε πληροφορίε στο ΣΥ. Εάν λοιπόν στη βάση δεδομένων δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι ξένοι μαχητέ από τι διάφορε χώρε, και τι να του κάνουμε που του ελέγχουμε. Σοβαρά τώρα. Ε, θα ενοχλήσετε τον κόσμο εκεί, ε, θα τους ελέγχετε και απλώς θα εκνευρίζετε και αν δεν μπορείτε να κάνετε διασταύρωση στοιχείων με μια βάση δεδομένων ε, για ποιοι μπορεί να είναι πιθανοί τρομοκράτες, άχρηστο θα είναι. Και επίσης θα φτιάξουμε ένα τμήμα αντιτρομοκρατικό στη Europol και πιο συγκεκριμένα θα είναι για τους ξένους μαχητές αλλά δεν προβλέπετε ότι οι τελωνιακοί υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών της Ευρωπόλ. Επομένως, για ποιο λόγο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα είναι ε, πολύ πιο επικριτικά. Αν διαβάζω το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ καλογραμμένο αλλά δεν προσφέρει καμία λύση. Δεν πρόκειται για διοικητικό. <coughs> Πρόβλημα είναι πολιτικό και τεχνικό. Συγγνώμη στους σοσιαλιστές. Εντάξει, δεχόμαστε τη συγγνώμη σα. Αναρωτιόμουν κι εγώ πού το πηγαίνατε. Χριστίνα. Ναι, πολλά ακούστηκαν και τα συμμερίζομαι. Όπως ότι πρέπει να είναι πολιτική η απόφαση. Το Σέγγεν είναι από τα θεμέλια της Ένωσης. Αρχίσαμε από ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και τελικά καταλήξαμε στο θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων αλλά και των ατόμων. Δεν θέλουμε βέβαια να επανέλθουμε σε μια απλή ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων. Τώρα θα ήθελα να επανέλθω σε δύο θέματα που δεν αναφέρθηκαν ακόμα και μένα αυτό με σοκάρει πολύ. Γίνεται λόγος για την Ουγγαρία και τον τείχο της, το τείχος της, τη φυλάκιση μεταναστών και άρα πρόκειται για παραβίαση ακόμα και της συνθήκης της Γενέβης. Πέρα και από το σεβασμό του ευρωπαϊκού δικαίου δεν γίνεται σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Λυπάμαι για την ψηφοφορία που έγινε στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα ενώ εμείς είχαμε καταθέσει τροπολογία για να χρησιμοποιηθεί επιτέλους το άρθρο 7 κατά της Ουγγαρίας και του κυρίου Ορμπάν γιατί η κράτηση μεταναστών είναι κάτι σκανδαλώδες. Πολλοί έχουμε ταραχτεί και το είπαμε στο Κοινοβούλιο και η Κομισιόν επίσης το απορρίπτει αυτό. Πρέπει όμως να εφαρμοστεί μια απλή αρχή. Όταν είναι κανείς στην Ένωση σέβεται τους κανόνες και τις συνθήκες. Άμα δεν τις σέβεται τότε γιατί να μείνει στην Ένωση. Και θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι τα άκρα. Όλοι οι ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα ως προς αυτά που γίνονται στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσα να μιλήσω και για τη Δανία αλλά δεν μιλάω. please. Κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς την Κομισιόν γιατί διαχώρισε ρητά μεταξύ Σέγγεν και των υπολείπων θεμάτων. Το πρόβλημα είναι το Δουβλίνο, όχι το Σέγγεν. Και ήρθε η στιγμή να δούμε πώς θα μπορούσε κανείς να οργανώσει αλλιώς τις αφήξεις στην Ευρώπη. Έγινε λόγος ας πούμε για ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Δυστυχώς αυτά ποτέ δεν ξεπέρασαν τις θεωρητικές ε, συζητήσεις. Εχθές ο Αντώνιο Γκουτιέρες είπε ότι πρέπει επιτέλους να δώσουμε μερικά χρήματα στις χώρες προέλευσης για να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί στα στρατόπεδα των προσφύγων. Και δεν είναι επομένω εκπληκτικό αφού δεν έγινε τίποτα ότι φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. η δική μου χώρα είναι χώρα διαμετακόμισης προσφύγων, περάσματος. Ε, και εμείς είχαμε δυσάρεστες εκπλήξεις διότι μερικοί από τους γείτονές μας άλλαξαν την πολιτική τους μονομερός και μείναμε με 5 εκατομμύρια ανθρώπους στα χέρια χάρηκα ιδιαίτερα που μπορέσαμε να λύσουμε λίγο πολύ αυτά τα προβλήματα με τη γειτονική μας χώρα την Γερμανία. Εγώ ζω σε μια συνοριακή περιοχή παραμεθόρια και βλέπω ότι είναι τεράστιοι οι αριθμοί των προσφύγων που καταφθάνουν. Μπορέσαμε να το διαχειριστούμε. Έχουμε 80.000 αιτητές ασύλου στην Αυστρία που θέλουν να παραμείνουν εκεί. Μπορεί να τους αναλάβει η χώρα ελπίζω. Αν και είναι ο ίδιος αριθμός με της Γερμανίας που είναι 10 φορές μεγαλύτερη. Δεν θα έπρεπε απλώς βέβαια να μεταφέρουμε τα προβλήματα της μίας χώρας στην άλλη. Πολλοί αρχικά ήταν υπέρ της επαναφοράς των ελέγχων στα σύνορα, αλλά κατάλαβαν ότι έχει αρνητικά αποτελέσματα. Στη δική μου περιφέρεια ας πούμε από τότε που καταργήθηκαν τα σύνορα αυξήθηκε η συνεργασία οικονομική και ξαφνικά δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία υγειονομικά επίσης γιατί η συνεργασία που υπήρχε και ιατρικά μεταξύ διάφορων παραμεθορίων νοσοκομείων ε, με την επαναφορά των ελέγχων δεν υπάρχει πια και αυτό είναι αρνητικό γενικά. Είναι πολύ σημαντικό να καταργηθούν αυτά τα σύνορα. Είδαμε ότι υπήρχαν ωφέλη στην πράξη. Το Σέγγεν ήταν τεράστια πρόοδος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τεράστιο και κτημένο, το οποίο δεν πρέπει να καταργήσουμε. Τώρα, ε, ερώτηση προς την Κομισιόν στο Στρασβούργο για δεύτερη φορά επιβλήθηκαν πολλοί έλεγχοι στα σύνορα. Ποιος είναι ο λόγος για αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε. Προσθέτω την κυρία Σπινέλη στον κατάλογο, λίγη εδώ ο κατάλογος, Κα Ναι. Μερικά ερωτήματα και σχόλια. Ερώτημα. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν αναφερθεί και αυτό είναι θέμα που χρόνια το συζητάμε και δεν έχει λυθεί. Βάλτε ακουστικά κυρία Κομίσιον. Σας ε, θέτει ερωτήματα η κυρία Σκά για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που είναι θέμα που το συζητάμε χρόνια από την προηγούμενη θητεία ζητούμε να μπει στο Σέγγεν η Ρουμανία και η Βουλγαρία από ό,τι ξέρουμε όμως δεν έχει γίνει τίποτα σχετικό για την ένταξη Ρουμανίας-Βουλγαρίας στο Σέγγεν πώς Πού, πού είναι τα πράγματα, υπάρχει, προβλέπετε ημερομηνία για τη Σουηδία. Θα ήθελα να γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται στα σύνορα. Τι συνοριακοί έλεγχοι γίνονται, έλεγχοι διαβατηρίων ή τίποτε άλλο. Τώρα για τους φράκτας. Υπάρχει κανένα πρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα, πότε θα καταργηθούν ε, τα σειρματοπλέγματα. Για το Σέγγεν μιλήσατε για τους λόγους για τους οποίους μπορεί να κλείνουν τα σύνορα των χωρών του Σέγγεν. Το κλείσιμο των συνόρων έχει χρησιμοποιηθεί ως πολιτική απειλή από διάφορες χώρες μέλη. Το έχετε πει αυτό δεν είμαι σίγουρη ότι είναι κάτι χρήσιμο, ούτε ότι είναι σοβαρός λόγος για κλείσιμο των συνόρων αυτός που αναφέρθηκε. Εφόσον οι χώρες μέλη όμως φαίνεται ότι θέλουν να επανέλθουν σε αυτό, πράγμα που είναι κατ' εμέ πρέπει παρόλα αυτά να καταλάβουν ότι χρησιμοποιήθηκε σαν απειλή από μερικές χώρες ενώ άλλες που δεν ήθελαν να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους για τις μετεγκαταστάσεις δεν συζητήθηκαν καθόλου. Πώς πήγαν οι συζητήσεις εκεί σχετικώς. Αν έχετε καμιά πληροφορία που μπορείτε να μας δώσετε θα ήμουν ευτυχής να την μάθω αναδολμές. συμφωνώ ότι η κύρια ευθύνη είναι των χωρών μιλών. Αλλά και η Κομισιόν έχει μια ευθύνη. Όπως επίσης είπαν άλλοι. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν θέλουμε υπαλληλική προσέγγιση αλλά πολιτική. Γιατί η Κομισιόν είναι ο κινητήρας της Ένωσης. Αν η Κομισιόν δεν αναλάβει την πολιτική της ευθύνη κατηγορώντας χώρες μέλη που παραβιάζουν τις δεσμεύσεις τους στην εφαρμογή του Σέγγεν τι θα γίνει γιατί αυτά είναι δικαιολογίες δίθεν καταπολέμησης της τραμακρατίας λοιπόν η Κομισιόν να μας τα πει αυτά και να αποδώσει ευθύνε. Είναι και αυτό δουλειά μας. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αφού δεν το κάνει η Επιτροπή αυτό. Εγώ τρομοκρατήθηκα την περασμένη εβδομάδα, εφρικίασα όταν ο κύριος Τίμερμανς που είναι και από την πολιτική μου οικογένεια ήρθε να μας εξηγήσει τη λογική αυτού του νέου, των νέων συνοριοφυλάκων. Και λέγοντας ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που θέλαμε, δηλαδή συνέχεια τρομοκρατία με πρόσφυγες. Δεν είμαι αφελής, δεν αγνοώ ότι μεταξύ των προσφύγων μπορεί να υπάρχουν τρομοκράτες που τους δίνετε ε, νέες ευκαιρίες, αλλά υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες που δεν αντιμετωπίζονται ούτε από τα κράτη-μέλη ούτε από την Κομισιόν. Και υπάρχουν επίσης αντιευρωπαϊστές που εκμεταλλεύονται αυτή τη σύγχυση. Ποτέ δεν θα υπάρξει πλήρης έλεγχος κάθε εκατοστού συνόρων, εξωτερικών συνόρων. Ποτέ. Μερικοί μιλάνε για θέλημα Θεού, αλλά αυτά είναι ανοησίες. Πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να τονίσει πρώτη ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης και διάσωσης του Σέγγεν, διότι το Σέγγεν είναι πολύ καλό εργαλείο, The problem. είναι να επενδύσουμε σε αυτά τα μέτρα όπως την ε, αέρια γέφυρα. Διότι οι άνθρωποι θα έρχονται ούτως ή άλλως. Και από την Πορτογαλία έρχονταν σε περιόδους όπου υπήρχαν παντού συνοριακοί έλεγχοι. Και κατάφερναν να πηγαίνουν οι άνθρωποι να εργαστούν σε άλλες χώρες. Θα συνεχίσει λοιπόν αυτό. Και τότε δεν προσπαθούσαν καν να σώσουν τη ζωή τους. Ήταν απλώς για βελτίωση. Αν τώρα λοιπόν θέλουμε να σώσουμε ζωές, των προσφύγων και των αιτητών ασύλου πρέπει να ξέρουμε ότι δεν θα πάψουν οι ροές. Γιατί να μην την οργανώσουμε καλύτερα λοιπόν με ασφαλέστερες διόδους και τρόπους καταγραφής ας πούμε. Εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να είναι στην πρωτοπορία να κάνει τέτοιες προτάσεις και δεν το βλέπω. τα επιχειρήματα των ακραίων δεξιών και αριστερών. Δεν εκμεταλλεύονται τους υπάρχοντες δρόμους και αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. ή αντιμετώπισης της καταπολέμησης της κερδοφορίας των δουλεμπόρων το λεγόμενο Golden Visa Program δεν το προσέχουν καθόλου. Αν ήμουν τρομοκράτησα θα ήξερα ότι είναι πολύ εύκολο να αγοράσει κανείς ηθαγένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι φρικιαστικό ότι συνεχίζει να το παραβλέπει η Κομισιόν αυτό. Συνδέονται τα προβλήματα για τους πλούσιους είναι ευκολότερο η απόκτηση ηθαγένειας από ό,τι για τους πτωχότερους. Τέλος ο κύριος Γκουτιέρες που τελειώνει τη, δεκαετή θητεία του ως ύπατος αρμοστής είπε ότι η αντίδρασή μας είναι ανεπαρκής και καθυστερημένη. Και αυτό ωφελεί τους ακραίους. που τολμάνε ακόμη και να κατάσχουν τα κοσμήματα των προσφύγων. Ευχαριστώ πολύ. Τέντερ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ακούγεται μια βοή εδώ στην αίθουσα. Πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση του μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λέμε ότι στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε η Κομισιόν να πει στα κράτη-μέλη τι δεν μπορούν να παραβιάσουν και ε, θέλουμε να γνωρίζουμε πέραν ε, του αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται διπλωματικά και με πολύ δύσκολες συνθήκες γιατί τα κράτη-μέλη έχουν ε, όλο ένα και περισσότερο εγωιστικά συμφέροντα, υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Μας διαλύουν τη Σέγγεν και μας διαλύουν την Ευρώπη και αυτό είναι ουσιώδες. Εμείς αναφερόμαστε σε ασφαλείς οδούς, σε ανθρωπιστική θεώρηση διαβατηρίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το σύστημα αποσυντήθεται γιατί δεν κάνουμε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των Ευρωπαίων και αυτό που είναι ανθρωπιστικά ε, λογικό για τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει ως Ευρωπαίοι. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει ποιες είναι οι διαχωριστικές γραμμές ε, τις οποίες δεν μπορούμε να υπερβούμε. Πρέπει να μας το πούνε, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει τη δουλειά τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζητόσκη. Ζητώ συγγνώμη στην Άννα αλλά πρέπει να κάνω το εξή σχόλιο. Ωραία και καλά που έχετε κάποιον από την Πορτογαλία να επικρίνει αυτές τις ε, χρυσές θεωρήσεις διαβατηρίων, της Golden Visa, αλλά δεν μπορώ να τα αφήσω να περάσει έτσι. Η Πορτογαλία μας άνοιξε το δρόμο για αυτές τις χρυσές θεωρήσεις. Να λέμε όμως και τα πράγματα με το όνομά τους. Η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Συμφωνώ με τον συνάδελφο τον κύριο Ντεπρέ και να σας πω ότι εχθές ήδη ε, η βάση δεδομένων ε, της Ευρωπόλ έχει 700 Ευρωπαίους συγγνώμη, 700.000 ξένους μαχητές και 5.000 εξ αυτών είναι στο Βέλγιο. Έχουμε δηλαδή 5.000 Βέλγους που ξέρουμε ότι έχουν πάει να πολεμήσουν για το Ισλαμικό κράτος για κάποιο χρόνο. Ε, η Γαλλία έχει αντίστοιχους αριθμούς, η Γερμανία ίσως λιγότερους. Να είμαστε λίγο ειλικρινές όμως. Ε, τι κάναμε εμεί τα τελευταίο χρόνο. Μπορεί να έχουμε τον εξαιρετικό χώρο Σέγγερ, μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά σύνορα και ελέγχου στα σύνορα, αλλά αν δεν ανταλλάζονται πληροφορίες, αν δεν εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον στην οικογένειά μας, δεν υπάρχει και κανένας λόγος να τα κάνουμε όλα αυτά. Ε, θέλετε μια πολιτική δήλωση, ορίστε. Αν αναφερόμαστε στο κεκτημένο Σέγγεν του χρόνου, θα ξανακάνω το ίδιο σχόλιο και θα μου λέτε και πάλι ότι έχουμε τη βάση δεδομένων που έχει 20.000 ονόματα. Πολύ ωραία. στα σύνορα μεταξύ Γαλλίας και Λουξεμβούργου έχει αστυνομικούς που ελέγχουν τα ταξιδιωτικό σας έγγραφα. Ε, μια ματιά ρίχνουν, τα γυρνάνε και απ' την άλλη, σας τα δίνουν και σας εύχονται καλό ταξίδι. Αυτό είναι τίποτα, παράσταση ε, και δεν θα αλλάξει και τίποτα. Ο τρομοκράτης Αν ο έλεγχος γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, αν δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, αν μας δείχνει ένα αυθεντικό διαβατήριο, ε, δεν έχει κανένα νόημα. Κατά την άποψή μου, η Σέγγεν είναι τα πάντα. Είναι η ελεύθερη κυκλοφορία. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από αυτό. Εγώ είμαι Τσέχος και θυμάμαι τις παλιές ημέρες που κοιτούσαμε τα φράχτες που μας απέκλαιαν από τη Γερμανία και από την Αυστρία και μας έλεγαν οι κομμουνιστές ηγέτες μας ότι, είμαστε μπροστά, ότι δεν είμαστε μπροστά από το φράχτη αλλά είμαστε πίσω από το φράχτη και το ξέραμε αυτό. Μόλις επέστρεψα από την Κούβα και σας συστήνω όλων να πάτε στην Κούβα και να δείτε πώς είναι η ζωή πίσω από το φράχτη. Επικρίνουμε την Ουγγαρία διότι πάντα βρίσκουμε έναν αποδιοπομπαίο τράγο και τα ρίχνουμε όλα σε αυτόν. Ε, πήγα στο Καλέ για να δω τι γίνεται και θα μπορούσα να επικρίνω πολύ κάλλιστα την κατάσταση εκεί. Και δεν νομίζω όμως ότι πρέπει απλώς να εξαπολύουμε κατηγορίες. Πρέπει να υποστηρίξουμε ένα τον άλλον και να δείξουμε ε, ε, παραδείγματα καλής πρακτικής. Δύο ακόμα πράγματα. Ξέρω ότι βιαζόμαστε. Ανθρωπιστικές θεωρήσεις διαβατηρίων. Συμφωνώ 100% με αυτό που ακούστηκε. Αλλά πόσες από αυτές τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις μπορούμε να δώσουμε. Πόσες ε, θα εκδώσουν οι κυβερνήσεις. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ε, είναι και αδιέξοδο. Το συζητάμε ένα χρόνο τώρα και θυμάμαι και κάποια από τις πρώτες σας ομιλίες όπου κάνατε τη συγκεκριμένη πρόταση τίποτα από εκεί και πέρα. Κενά λόγια και δεν συνέβη τίποτα. Πρέπει να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο, αλλιώς θα μείνουν όλα κενό γράμμα. Και δεν θα κάνω και την τελευταία μου παρατήρηση γιατί ούτως ή άλλως τέσσερα λεπτά σας μιλάω χωρίς διακοπή. Τελευταία μιλήτρια η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ανησυχώ κι εγώ πάρα πολύ. διότι διαχέονται αυτές οι πολιτικές κλειστών συνόρων. Ήδη 8 χώρες έχουν επαναφέρει ελέγχους και επίσης ανησυχώ και με την ευκολία με την οποία το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζουν να εξαπολύουν απειλές ε, για αποκλεισμό από τη Σέγγεν αν τα hot spot δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Υπάρχει κάτι επιπλέον όμως που με ανησυχεί. Δεν θα ήθελα να επικεντρωθούμε μόνο στο κλείσιμο των συνόρων, αλλά και στην επιλογή που γίνεται από κάποιες κυβερνήσεις, είτε της Ένωσης, είτε ε, καθοδόν προς την Ένωση, την επιλογή κατά συγκεκριμένων ε, υπηκών από κάποιες χώρες και την θρησκεία τους. Θεωρώ ότι είναι πολύ ανησυχητικό αυτό ε, για τα όσα συμβαίνουν σε αυτή την οδό από τα Βαλκάνια και εδώ συμφωνώ και με την Άννα Γκόμες. Η ευθύνη είναι σίγουρα των κρατών μελών αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων, επομένως και του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, άρα έχει και κάποιες συγκεκριμένες ευθύνες. Αδιαμφισβήτητες. Κάτι τελευταίο, το οποίο θα ήθελα να πω στη συνάδελφο Κοράτσα Μπίλτ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με διορθώσατε. Εγώ αναφέρθηκα στο συνταγματικό δικαστήριο στη Σουηδία, το οποίο ε, κατήγγειλε τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης, πρόκειται όμως για ένα συμβούλιο το οποίο είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Έκανα το λάθος διότι το συμβούλιο αυτό ελέγχει, εξαρτάται μένα από την κυβέρνηση, αλλά ελέγχει την εγκυρότητα της νομοθεσίας, που σε, κάτι που σε πολλές χώρες είναι αρμοδιότητα του συνταγματικού δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, επ' αυτού για τη συζήτηση αυτή. Όλοι αναφερθήκατε στο θέμα αυτό και με πάθος αλλά και με πολύ τεχνική γνώση. Ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. πριν τα θέσουμε όλα αυτά ή μάλλον τα αποθέσουμε όλα αυτά στους ώμους ενός διευθυντού τμήματος όπως είναι εδώ ο παριστάμενος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσουμε και στη βάση των εκθέσεων αξιολόγησης που διαθέτουμε. Αυτά μας τα αναθέτει ως αρμοδιότητα και το άρθρο 70 της συνθήκης. Και αυτά θα τα φροντίσουν οι συντονιστές την επόμενη χρονιά. Το ΑΔΕ άρθρο 17 λέει ότι ορισμένες εκθέσεις αξιολογήσεων πρέπει να καθίστανται δημόσιο κτήμα. Ο κ. Κόιστερ να το θίξει το θέμα αυτό στην απάντησή του. Πάντως, σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις ε, εξαιρετικά στις παρεμβάσεις σας. Κύριε Δεκόιστερ, κάνετε προσπάθεια να απαντήσετε. Αντιλαμβάνομαι βέβαια πόσο σημαντική είναι η πολιτική διάσταση του θέματος. Κάντε ό,τι μπορείτε. Και βεβαίως γνωρίζετε η κατάσταση αυτή έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα, είναι όμως και μια διαρκής ε, ε, εξέλιξη αυτή στα μάτια μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. αντιλήφθη το πολιτικό μήνυμα και θα το διαβιβάσω στα πολιτικά αφεντικά μου. Τώρα για τα διάφορα θέματα, πολυπληθή άλλωστε που θέσατε, θα προσπαθήσω να τα ομαδοποιήσω. Πρώτο, για το νέο μηχανισμό αξιολογήσεως Schengen και τις κυβερνήσεις. Οι εκθέσεις που γίνονται μετά από τις επισκέψεις διαβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. είναι βέβαια περιορισμένης χρήσεως, έχουν μια διαβάθμιση, δίνονται λοιπόν στη γραμματεία της Επιτροπής σας. Και αν τα μέλη σας χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούμε να τους διαθέσουμε. Απόλυτη διαθεσιμότητα εκ μέρους μας να προχωρήσουμε σε τέτοιες συζητήσεις μαζί σας. Για τους φράχτες τώρα. Μία βουλευτή σας ανέφερε την παραδοσιακή θέση ας πούμε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους φράχτες. Βεβαίω, το τι είδους εποπτεία των συνόρων θα κάνουν οι χώρες μέλη είναι δική τους υπόθεση. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπέρ των φραχτών, Όταν πάντως μια χώρα εγείρει ένα φράχτη, πρέπει να σεβαστεί την αρχή του νόμου ρεφουλμών, Δηλαδή, όσοι προσέρχονται εκεί θα πρέπει να μπορούν να καταθέσουν αίτηση ασύλου. Η χρήση συνόρων τώρα σε εσωτερικά σύνορα είναι ακόμα πιο ευαίσθητο θέμα. Διότι καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης Schengen τα εσωτερικά σύνορα μπορούν να τα διέρχονται οι ενδιαφερόμενοι οπουδήποτε. Το να δει λοιπόν εκεί μια υποδομή που συνίσταται σε φράχτες όταν επαναφέρονται οι εσωτερικοί συνορικοί έλεγχοι μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβαίνει το κεκτημένο του Σέγγεν και το πνεύμα του. Από την άλλη μεριά το είδαμε αυτό και στα σύνορα μεταξύ Σλοβενίας και Αυστρίας όπου ανηγέθηκαν προσωρινοί φράχτες περισσότερο για να κατευθύνουν τις ροές των, μεταναστών έτσι ώστε να γίνεται η μετακίνησή τους με κάποια τάξη. Για τα σχόλια που έγιναν τώρα από ορισμένου ευρωβουλευτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της είπατε ως θεματοφύλαξη των συνθήκων Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Αυτό κάνουμε. Εξετάζουμε την κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται και στην Ουγγαρία και στις άλλες χώρες. Εξετάζουμε τι κάνει η Ελλάδα και για την εφαρμογή του Σέγγεν και του κεκτημένου για το άσυλο. Ακολουθούμε την οδό αυτή. Να γνωρίζετε επίσης ότι οι διαδικασίες προσφυγής Χρειάζεται πολύ χρόνο συνήθω. Αν χρειαστεί κάποια φορά να πάμε στο δικαστήριο, είναι θέμα, όπως είπα, μιας χρονοβόρας διαδικασίας. Εκ παραλλήλου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί και μια άλλη προσέγγιση, δηλαδή προσπαθεί να συμβάλλει στην εφαρμογή του κεκτημένου επιτόπου. Για παράδειγμα, για τα hot spot, η ομάδα έχει ομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει ομάδες για να συντονίζουν το έργο των διαφόρων οργανισμών, των τοπικών αρχών κλπ. για να βελτιωθεί η κατάσταση. Συμβάλλοντας έτσι σε ορθότερη εφαρμογή του κεκτημένου ασύλου και Σέγγεν. Δεν είναι δηλαδή να προτιμήσουμε ή τη μια ή την άλλη προσέγγιση, μπορούν να ακολουθούνται και δυο εκ παραλίδου. Τώρα, η ανθρωπιστική βίζα. Γνωρίζετε ότι αυτό εκπίπτει την αρμοδιοτήτων μου. Θα το αφήσω αυτό για τις αρμόδιε συναδέλφου. Να πείτε όμως ότι η Κομισιόν δεν κάνει τίποτε, δεν συμφωνώ απόλυτα. Μερικοί την λένε ανθρωπιστική βίζα, υπάρχει και η μετεγκατάσταση. Και στη μετεγκατάσταση έκανε προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι άνθρωποι που επωφελούνται από τη μετεγκατάσταση δεν λαμβάνουν ανθρωπιστική ή άλλου είδου βίζα, όμως μπαίνουν στη διαδικασία της μετεγκατάστασης. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν γίνονται κάποια πράγματα. Ίσως να μην είναι επαρκή, ίσως τα νούμερα να μην είναι αρκετά υψηλά. Αλλά και αυτό είναι πιο πολύ πολιτική συζήτηση. Μιλήσατε και για την διάρκεια των προσωρινών ελέγχων. Δύο μήνες και έξι μήνες είναι τα χρονικά όρια που ισχύουν όταν μονομερώς προχωρούν σε επανεισαγωγή ελέγχων οι χώρες μέλη. Για ορισμένους λόγους προβλέπονται ρητά. Τα δύο χρόνια που ανέφερα εγώ εφαρμόζεται σε μια πολύ ειδική περίπτωση όταν έχει γίνει η αξιολόγηση Σέγγεν και όταν έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ελλείψεις στην εφαρμογή του κεκτημένου για τα εξωτερικά σύνορα και όταν η οικία χώρα μέρος δεν λαμβάνει άμεσα μέτρα. Τότε μπορεί να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο να επιτρέψει στις χώρες μέλη να επανεισαγάγουν ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Εάν η μη ανάληψη δράσης όντως επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν Εκεί αρχίζει από 6 μήνες και το ανώτατο όριο της συνολικής περίοδου μπορεί να φτάσει στα 2 χρόνια. Σχετικά με τους αστυνομικούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Ορισμένες χώρες μέλη προσέφυγαν στην safeguard clause και αναφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλες χώρες μέλη κάνουν αστυνομικού ελέγχου που μπορούν να εφαρμόζονται σύμφωνα με το κεκτημένο Σέγγεν ακόμα και σε περιοχές εγγύς των εσωτερικών συνόρων. Μια συζήτηση που έχει γίνει και πολλές φορές άλλωστε. Πότε δηλαδή οι αστυνομικοί έλεγχοι συνιστούν στην πραγματικότητα συνοριακού ελέγχου, Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση. Τώρα για τους αλλοδαπούς σοσιαλιστές μαχητές. Αυτή η συζήτηση γίνει όταν θα μιλήσουμε για τη στοχευμένη πρόταση για τα σύνορα και ποιες βάσεις δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν. Δεν θα καταστήσει αυτό αδύνατη την μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών. μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά όταν θα έρθουμε στη συζήτηση εκείνη τη Έγιναν και μερικέ ερωτήσει για Βουλγαρία-Ρουμανία. Για αυτό το θέμα δεν γνωρίζω αν έχει γίνει καμία πρόοδος πρόσφατα. Ε, ούτε μπορώ να σας πληροφορήσω άρα. Δεν είμαι σίγουρος καν ότι έχει συζητηθεί πρόσφατα γιατί μια επέκταση του Σέγγεν δεν την εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Πρώτα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα που συζητήσαμε σήμερα και μετά να δούμε αν χρειαστεί επέκταση ή διεύρυνση του Σέγγεν. Τώρα, όσο στο τι κάνουν οι χώρες μέλη όταν επανεισάγουν, αναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους, <clears throat> θα ήθελα να σας αναφέρω τα επιστολάς που έστειλε που στέλνει η Κομισιόν στο Κοινοβούλιο κάθε φορά που μια χώρα μέλος μας γνωστοποιεί την επαναφορά. Ας πούμε, που, ποια είναι τα σημεία εισόδου, τι έλεγχοι επιβάλλονται κτλ. Αυτά συστηματικά στέλνονται στο Κοινοβούλιο και περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα ανέφερα όλα, μπορεί να παρέβλεψα τίποτε, αλλά εγώ χρειάζομαι διακοπές. Ναι, άνθρωπος είστε και εσείς φαίνεται. Είχα πει από την αρχή ότι το θέμα του Σέγγεν είναι τόσο τεράστιο ώστε δεν περιμέναμε να μας δώσετε θαύματα να μας προτείνετε. Απλώς υπό το 70 έχουμε και εμείς ευθύνες και έχουν ακουστεί πολλά και έντονα. Τον Ιανουάριο λοιπόν θα γίνει μια έκτακτη συνεδρίασή μας με, για τις αξιολογήσεις πρώτα αν οι συντονιστές το εγκρίνουν. στην πρώτη μας συνεδρίαση του Ιανουαρίου. Για να μην χάσουμε την ορμή λοιπόν από αυτή την εξαιρετική συζήτηση, την τελευταία αυτή μέρα πριν από τα χρήση Χριστούγεννα, πόσο σκληρά δουλεύει η Επιτροπή μας, το θαυμάζω, σας κατευχαριστώ. Φυσικά και εσείς κύριοι εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορείτε να πάτε διακοπές αλλά να μην ξαναγράψετε πράγματα κατά των σοσιαλιστών στα σύνορα. Τώρα, αν μείνει κανείς, έχουμε ακόμη μια έκθεση και μερικά άλλα θέματα. Το σημείο 9. Εξασφάλιση κοινού υψηλού επίπεδου ασφαλεία δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου του Γιάνν Άλμπρεχτ. Αν θέλεις Γιάνν να μας κάνεις μια σύντομη ενημέρωση, η πρόταση οδηγίας για το κτλ. Επαναλαμβάνω για την εξασφάλιση κοινού επίπεδου ασφαλείας, διεκτήμων και πληροφοριών από ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει το λόγο. Σας κατευχαριστώ όλους εσάς που μείνατε μέχρι τώρα για να μιλήσουμε για τα τελευταία αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την οδηγία ασφαλείας στο δίκτυο εισηγητής ο Ανδρέας Σβάμπ. Εγώ είμαι συντάξη χρηματοδότησης για την Λίμπε και Σκιώδη ΣΥΜΚΟ. Είναι καλό και σωστό που τελειώσαμε την εξέταση αυτής της οδηγίας τώρα. Χρειάστηκε χρόνος βέβαια. Και αυτό δεν οφείλεται, η καθυστέρηση δεν οφείλεται στο κοινοβούλιο αλλά στα κράτη-μέλη και την έλλειψη θέλησής τους να μοιραστούν πληροφορίες. Το ίδιο πρόβλημα νομίζω έχουμε εδώ όπως και μετά αστυνομικά θέματα και γενικά της ασφάλειας των πληροφοριών. Πολύ συχνά λείπει η θέληση αλλά και η εμπιστοσύνη για την χορήγηση πληροφοριών σε θέματα ασφαλείας, ηλεκτρονικής ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά Πρόκειται για την πρώτη συνδυασμένη προσπάθεια βελτίωσης της ασφάλειας στην Ένωση σε αυτά τα θέματα. Η έλλειψη θέλησης νομίζω σημαίνει ότι στο μέλλον μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα και θα χρειαστεί να γίνουν. Ιδιαίτερα σε τομείς και θέματα όπου που δεν είναι τόσο περιορισμένα όπως εδώ αλλά οι ζωτικές υποδομές και η χρήση όλων των σχετικών τεχνολογιών. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό αργότερα στο χρόνο. Αλλά όπως είπα είναι η πρώτη συνδυασμένη προσπάθεια δημιουργίας ενός ελαχίστου επίπεδου ηλεκτρονικής ασφαλείας τουλάχιστον για ζωτικέ υποδομές. Για την Επιτροπή μας ένα ήταν το κύριο θέμα στις διαπραγματεύσεις αυτές ή μάλλον δύο. Ένα θέμα δηλαδή δύο. Και αυτό τα δύο θέματα ήταν ένα ο σεβασμός του κεκτημένου για τα προσωπικά δεδομένα Αυτό έγινε. Και το δεύτερο αν υπάρχει παραβίαση ασφαλείας κάπου να πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση. Τώρα προβλέπετε ότι πρέπει να γνωστοποιείται ή παραβίαση ασφαλείας κάπου, αλλά βέβαια και αν τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων, πάλι να γίνεται γνωστοποίηση. Για να είναι βέβαιο ότι οι αρχές που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των δεδομένων θα το γνωρίζουν. Και αυτό έγινε. Είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι και από την Επιτροπή μας απλώς Ένα τελευταίο που πρέπει να ξέρετε, σε σύγκριση με την αρχή των διαπραγματεύσεων και την πρώτη πρόταση της Κομισιόν, τώρα υπάρχουν πρότυπα και για τους προμηθευτές χορηγητές των ε, υπηρεσιών. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δηλαδή γνωρίζουν τώρα ότι μπορεί να χρειαστεί να τους εξετάσουμε και αυτούς αλλά με διαφορετική προσέγγιση. Το γενικό επίπεδο προστασίας στην οδηγία αυτή προβλέπει μία ελάχιστη εναρμόνιση ενώ για τους προμηθευτάς maximum επίπεδο. Γιατί το επίπεδο προστασίας εκείνο τον τομέα δεν είναι πολύ ψηλό και πρέπει να ληφθεί υπόψη και για την περαιτέρω αναθεώρηση για να υπάρξει εξισορρόπηση. Τέλος, για το χρονοδιάγραμμα. Η έγκριση στην ΙΜΚΟ προβλέπεται για τις 14 Ιανουαρίου, οπότε και θα γίνει η ανακοίνωση στην όλο. Ολομέλεια κάποτε αργότερα, θέση ενισχύει 27 μήνες μετά τη δημοσίευση της οδηγίας νης στη δημιουργήσιμη εφημερίδα. Νομίζω θα χρειαστεί πολύ χρόνος και για τις γλωσσικές επαληθεύσεις. Δεν ξέρω πότε θα φτάσει στην Ολομέλεια, αλλά κάποτε την άνοιξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ε, ήταν πολύ σημαντική η δουλειά αυτή μεταξύ ημών και της Επιτροπής ΥΜΚΟ και νομίζω ότι κάποια από τα θέματα τα οποία προέκυψαν κυρίως για την ε, ιδιωτική ζωή οργανώθηκαν τόσο πολλά στην Επιτροπή μας πριν από μερικές εβδομάδες και επειδή είναι τόσες πολλές ε, οι εξελίξεις πολλοί δεν μπόρεσαν να παραστούν ο κύριος ε, Μπόνι ε, ασχολείται και με τα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά για την Επιτροπή μας και αρκετά χρονοβόρα. Χαίρομαι λοιπόν, διότι πρόκειται για κρίσιμους τομείς ε, για μας και επηρεάζουν φυσικά και την ΙΜΚΟ με διάφορους τρόπους. Θέλει κανείς να πει κάτι? Αν όχι, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο και να περάσουμε στο πρώτο τελευταίο σημείο που είναι η έκθεση της Επιτροπής ε, που αξιολογεί την κατάσταση της μη αμοιβαιότητας με κάποιες ε, τρίτες χώρες στον τομέα της πολιτικής θεωρήσεων ε, διαβατηρίων. Είναι τμήμα του λεγόμενου μηχανισμού αμοιβαιότητας που διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τα ίδια δικαιώματα και απαλλάσσονται από θεώρηση διαβατηρίων από τρίτες χώρες. Έχουμε κάποια στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναστολή της απαλλαγής θεωρήσεων για υπηκόους τρίτων χωρών όπου η κατάσταση δεν την χάνει πλήρους αμοιβαιότητας. Υπάρχουν δύο προηγούμενε εκθέσει Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν αξιολόγηση των κοινοποιήσεων από τα κρατη κατά τη Αυστραλία, του Μπρουνέη, του Ντάρελ Σαλάμ, τη ε, ε, του Καναδά, τη Ιαπωνία και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην τρίτη έκθεση περιγράφονται συγκεκριμένα βήματα ε, τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν από συγκεκριμένε χώρε και καμία από τι χώρε αυτέ δεν ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαλλαγή από τη θεώρηση διαβατηρίων και γι' αυτό ακριβώς ε, δεν έχει ανασταλεί η απαλλαγή. πρέπει να σας πω ότι συζητήθηκε και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, συζητήθηκαν αλλαγές το πρόγραμμα απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων ε, για λόγω των τρομικροτικών επιθέσεων. Παραδείγματο χάρη ότι οι ανθρώπου που έχουν επισκεφθεί το Ιράκ και το Αφγανιστάν θα χρειάζεται θεώρηση διαβατηρίων για να επισκεφθούν και επομένω αυτή είναι περίπτωση μια αμοιβαιότητα. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στου εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα ενημερώσουν για όλε αυτέ τι εξελίξει και από εκεί και πέρα θα έχουν το λόγο τα μέλη. Από την Κομισιόν Έχουμε τον αρμόδιο ναι. εκπρόσωπο. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είμαι εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε εδώ το Σεπτέμβριο για να σας αναφέρει την κατάσταση περί αμοιβαιότητα ημί. και έκτοτε έχουμε εκδώσει και την τρίτη μας έκθεση και όπως είπατε μας ανησυχούν και εξελίξεις στις Ηνωμένες θα ήθελα λοιπόν να σας πω λίγο που βρισκόμαστε. Θα ξεκινήσω με την έκθεση και θα ανακεφαλίσω λίγο πώς λειτουργεί ο μηχανισμός αμοιβαιότητας. Όπως είπατε, ε, σε πρώτο στάδιο κάθε έξι μήνες είτε πρέπει να εγκρίνονται προσωρινά μέτρα, δηλαδή αναστολή της απαλλαγής διαβατηρίων ή απλώς να γίνεται μια έκθεση της κατάστασης. Έχουμε υποβάλει την τρίτη μας έκθεση, υπευλήθη στις 5 Νοεμβρίου και δεν έχουμε εγκρίνει κάποια μέτρα για, τις, ε, για αναστολή. Ε, το επόμενο στάδιο του μηχανισμού προβλέπει ότι αν υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις μη αμοιβαιότητας στις 12 Απριλίου του 2016, δηλαδή δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης ε, της κοινοποίησης μη αμοιβαιότητας που ελήφθη από τα κράτη-μέλη, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει μέσω πράξης κατεξουσιοδότηση ε, μέτρα για προσωρινή αναστολή για 12 μήνες για υπηκόους τρίτων χωρών, ε, των χωρών που αφορά η μη αμοιβαιότητα. Σε λίγους μήνες λοιπόν θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Όπως ε, είπατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρεις εκθέσεις για την αναστολή επειδή υπάρχει συνεχής δέσμευση των ε, εν λόγω χωρών ε, για συζητήσεις και επειδή κανένα κράτος μέλος δεν μας ζήτησε να εγκρίνουμε προσωρινά μέτρα. Να σας πω λίγο πως έχει κατάσταση για κάθε μία από τις χώρες που αναφέρατε. Για την Αυστραλία καταρχάς. Η Αυστραλία ε, ήρε την απέτηση και για τη Ρουμανία και για την Κροατία ε, για διαμετακόμιση. Επομένως όσον αφορά την Αυστραλία θεωρούμε ότι υπάρχει πλήρης αμοιβαιότητα στα πλαίσια του μηχανισμού αμοιβαιότητας. Άρα η Αυστραλία είναι εντάξει. Μπρουνέι. Το Μπρουνέι είναι την απέτηση ε, για θεώρηση από, για την Κροατία, μας το κοινοποίησε, αλλά δεν εφαρμόζεται πλήρως. Ήρθαμε σε επαφή με την ε, αποστολή του Μπρουνέι και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, ε, και την αντιπροσωπεία στο Μπρουνέι και μας διαβίβασαν το ίδιο μήμενα. Το Μπρουνέι πρόσφατα ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η απαλλαγή θεώρησης διαβατηρίων για την Κροατία και παράταση από τις 14 στις 90 μέρες για το Λίχτενστάιν θα ξεκινήσει από 1η Πρώτου του 2016. Για αμοιβαιότητα λοιπόν για τον Μπρουνέι λογικά από 1η Πρώτου του 2016 θα έχουμε απαλλαγή οπότε είναι εντάξει και τον Μπρουνέι. Καναδάς. Οι υπηκόοι Βουλγαρίας και Ρουμανία χρειάζονται ακόμα θεώρηση διαβατηρίου για να ταξιδέψουν στον Καναδά και το πιο σημαντικό κριτήριο το οποίο εφαρμόζει ο Καναδά είναι η παραβίαση του ποσοστού μετανέσταση και το ποσοστό άρνησης θεωρήσεων. Τα ποσοστά είναι άνω του ε, ο κατοφλίου του 3% ε, που τίθεται τα τελευταία χρόνια και για τις δύο χώρες είναι πάνω από 17% και πάνω από 16% για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία αντίστοιχα. Μετά από αυτή την εισαγωγή από τον Καναδά του ηλεκτρονικού, της ηλεκτρονικής έγκρισης ε, ε, ε, από το Μάρτιο του 2016 για θεώρηση διαβατηρίου, ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα την επεκτείνει και για τους υπηκόους Βουλγαρίας και Ρουμανίας που ταξιδεύουν ε, που ταξίδευσαν, συγγνώμη, στον Καναδά με θεώρηση διαβατηρίου για τα τελευταία 10 χρόνια ή έχουν μια έγκυρη θεώρηση διαβατηρίου ΗΠΑ. Για αυτού τους ταξιδιώτες λοιπόν αυτό θα θεωρείται απαλλαγή θεώρηση. Επικροτούμε τη συγκεκριμένη πρόοδο, αλλά ο στόχο είναι να έχουμε απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων ανεφόρων για όλου του υπηκόου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των υπηκόων Βουλγαρια και Ρουμανία. Για την Βουλγαρία και τη Ρουμανία βέβαια ε, φαίνεται απίθανο μέχρι τον Απρίλιο του 2016 να υπάρχει πλήρης απαλλαγή διαβατηρίων. Η Ιαπωνία. Είχαμε θετικές εξελίξεις από την έκρηση της έκθεσης τον Νοέμβριο. Η Ιαπωνία κοινοποίησε στη Ρουμανία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεσή της να επεκτείνει την απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων και στη Ρουμανία. Ε, θα έλεγε κανονικά το 2015 αλλά θα παρατείνεται και για το 2016. Καλύπτει και ε, για προσωρινά διαβατήρια Ρουμανίας που δεν είναι βιομετρικά, ε, κάτι το οποίο που θα έχουν κοινοποιηθεί από τη Ρουμανία. Τώρα, πέντε κράτη-μέλη χρειάζονται θεώρηση διαβατηρίου για να πάνε στις ΗΠΑ. Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Πολωνία και Ρουμανία. Και εδώ δεν αναμένονται αλλαγέ μέχρι τον Απρίλιο του 2016. Το βασικό πρόβλημα είναι το ποσοστό άρνηση θεωρήσεων που είναι υψηλότερο για όλα αυτά τα κράτη-μέλη από το 3% που ε, καθορίζεται στην νομοθεσία των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση είπαμε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το πρόγραμμα απαλλαγή θεωρήσεων διαβατηρίων και για άλλους Ευρωπαίους πολίτες και έχουν υπάρξει περαιτέρω εξελίξεις όπως αναφέρεται. Ήδη από τέλη Νοεμβρίου ο Λευκός Οίκο ανακοίνωσε μία σειρά από αλλαγέ που σχετίζονται με την ασφάλεια για το πρόγραμμα απαλλαγή θεωρήσεων και τα πιο σημαντικά είναι τα εξή. Συλλογή πληροφοριών από ταξιδιώτες ε, για οποιαδήποτε ταξίδια ε, σε χώρες οι οποίες ε, για τις Ηνωμένε Πολιτείε αποτελούν ε, ασφαλή λιμένα για τρομοκράτες, δηλαδή Συρία και Ιράκ και θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη αίτηση με αυτή του ΕΣΤΕ. Θέλω να εξετάσουν και τη δυνατότητα ενός πιλωτικού προγράμματος για να συλλέγει βιομετρικά στοιχεία, δακτυλικά αποτυπώμενα και φωτογραφίες για τους ταξιδιώτες της απαλλαγής θεωρήσεων ευατηρίων και επίσης θα επανεξετάσουν τις χώρες και θα ε, πρέπει επιμένουν από αυτές τις χώρες να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες ε, και για πιθανούς τρομοκράτες και θέλουν να ενισχύσουν και τον έλεγχο των συνόρων και να επιμείνουν ότι όλες οι χώρες που βρίσκονται στα προγράμματα ε, απαλλαγής θεωρήσεων θα πρέπει να ελέγχουν πρόσφυγες και τυχόν ύποπτους τρομοκράτες. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο Μίλλερ, το οποίο απαιτεί να υπάρχουν βιομετρικά διαβατήρια για όλους τους ταξιδιώτες, ε, πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας ε, PNR, ε, εκτεταμένη χρήση βάσεων δεδομένων της Ευρωπόλ και να αναφέρονται και στοιχεία για τυχόν κλαπέντα διαβατήρια. Αυτό θα αποκλείει και ταξιδιώτες που τα τελευταία πέντε χρόνια επισκέφθηκαν τη Συρία, το Ιράν, το Ιράκ και το Σουδάν. Επομένως περισσότερες χώρες από αυτές που αναφέρονταν ή οποιαδήποτε άλλη χώρα ε, που αποφασίζει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι θεωρείται ύποπτη ε, ή ε, πολίτες με μεικτή υπηκότητα, παραδείγματος χάρη γαλλοσύρο υπήκο. Την περασμένη εβδομάδα το νομοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε και από τη Γερουσία και από το Κογκρέσο και μάλλον συγγνώμη ένα άλλο νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει την ίδια διατύπωση με το νομοσχέδιο Μίλλερ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της προς τις ΗΠΑ για αυτές τις διατάξεις και είπαν ότι θα επηρεάσουν αρνητικά τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν καλή την πίστη στις χώρες αυτές, παραδείγματος χάρη επιχειρηματίες που έχουν ε, σκοπούς επιχειρήσεων ή ε, υπηκόους με διτή υπηκότητα. Ε, είναι πολύ δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί μάλιστα αυτό στην πράξη, πώς μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες ότι υπήρξαν ταξίδια προς τις χώρες αυτές και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εξήγησε και στους εταίρους της από τις ΗΠΑ τι έχει ήδη γίνει σε θέματα ασφαλείας σε διάφορους τομείς, παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό PNR, την Οδηγία για την Τρομοκρατία, τη Δέσμη Μέτρων για τα Σύνορα, για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη ριζοσπαστικοποίηση. Είπαμε ότι αντί να ε, δυσκολεύουμε ταξιδιώτες ε, που ταξιδεύουν καλή την πίστη, θα πρέπει να βελτιώσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών για συγκεκριμένες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη τρομοκράτες μαχητές, με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και επίσης επισημάναμε ότι πρέπει να εγκρίνουμε την, ε, να εγκρίνει συγγνώμη, το, η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών την νομοθεσία ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Παρά τις προσπάθειές μας και στις Ηνωμένε Πολιτείε και κατά τη συνάντηση με τον Πίτρο Παυραμόπουλο και τον ε, ε Υπουργό Ιστορικών Υποθέσεων των πολιτείων εγκρίθηκε σχετική νομοθεσία. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν άλλες μονομερείς δράσεις των πολιτείων πριν γίνουν επίσημες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, προσπαθεί συνεχώς να έχει επαφές ε, με το Υπουργείο Εσωτερικών, ε, Εσωτερικής Ασφάλειας για αυτό το νομοσχέδιο Omnibus. Νομίζω λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχει πλήρης αμεβαιότητα στις 12 Απριλίου του 2016 για τις Ηνωμένε Πολιτείες. Νομίζω ότι η κατάσταση μάλλον επιδεινώθηκε ε, και είναι πολύ πιο περίπλοκη. Όπω ξέρετε, ο μηχανισμό αμοιβαιότητα απαιτεί να εγκρίνουμε πράξη εξουσιοδότηση αν μέχρι τι 12 Απριλίου του 2016 η τρίτη χώρα δεν έχει άρει την απέτηση για απαλλαγή θεώρηση διαβατηρίου. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Ξέρω ότι υπάρχει και έκθεση από τη νομική υπηρεσία για μια δικαστική υπόθεση ε, για το κατά πόσο θα πρέπει να γίνεται με πράξη εξουσιοδότηση, με εκτελεστική πράξη, αλλά εμεί βάσει δικαίου πρέπει να ζητήσουμε πράξη κατεξουσιοδότηση. Εάν η πράξη εξουσιοδότηση εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή, εάν δεν υπάρχει ένσταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο εντό τεσσάρων μηνών ε, από την κοινοποίησή τη, θα ξεκινήσει η εφαρμογή τη. Δεν θα αρχίσω τι εικασίε τώρα για το χρονοδιάγραμμα τη ε, υποβολή τη πράξη εξουσιοδότηση. Πρέπει από τι 12 Απριλίου του 2016 να αξιολογήσουμε την κατάσταση, αλλά σα διαβεβαιώ ότι θα γίνει σεβαστή η συνεννόηση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πράξεις εξουσιοδότηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Σα ευχαριστώ πολύ. Μία μόνο αίτηση λήψη του λόγου από τον κύριο... Ευχαριστώ. Χάλαχα Θα ήθελα να βεβαιωθώ ότι όσοι έχουν την ηθαγένεια ή υπηκότητα μίας από τις ενωσιακές χώρες εννοείται όταν μιλάτε για dual citizenship και όχι τη Συρίας και τέτοια. Ναι, όσοι εκτός από ενωσιακή ηθαγένεια έχουν και ηθαγένεια Συρίας, Ιράν, Ιράκ ή Σουδάν. Αν και το νομοσχέδιο επίσης προβλέπει να προσθεθούν ίσως και άλλες χώρες. Αν δεν έχετε τίποτε άλλο, νομίζω το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε με τους συντονιστές πλέον για να συζητήσουμε ε, τι δράση θα αναλάβουμε εκ μέρους μας για την... Ε, εν μιλώ για τη συνάντηση του Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη του θέματος και έρχομαι στο επόμενο θέμα. Φτάνουμε σχεδόν στο 11. Πρώτα πρόκειται για την απόφαση του δικαστηριού της 16 Ιουλίου 2015 για την ε, ακύρωση των αθεωρημένων μηχανισμού αμοιβαιότητας. και για τη μερική ακύρωση κανονισμού του 2013. Πρόκειται για κατεξουσιοδότηση πράξης για δαπάνες για κοστή των χωρών και εκεί το δικαστήριο απεφάνθη ότι για τις κατεξουσιοδότησης πράξης και τα λοιπά. Και να, δώσει, να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ για την ευγενή σας πρόσκληση να σας αναπτύξω το θέμα ο εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας. Δεν το κάναμε επίτηδες να σας δώσουμε το λόγο στην τελευταία συνεδρίαση. Θα είμαι σύντομος, λέει ο εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας, δεν θα επαναλάβω, δεν θα εξηγήσω ολόκληρο το πλαίσιο. Θα θυμάστε ότι προδιετίας είχε εγκριθεί το κείμενο το, κατά το οποίο έγινε η προσφυγή τώρα και οι συνάδελφοί μου της ε, DG Home εξήγησαν αυτή τη διαδικασία τριών σταδίων στην αρχή της οποίας εάν μία από τις τρίτες χώρες που έχει ε, απολαύσει την απαλλαγή από προξενικές θεωρίες αν τις επαναφέρει δηλαδή για τους ε, ε, ε υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατηρηθεί το καθεστώς αυτό, τότε η αναστολή λαμβάνει τη μορφή τροποποίησης του παρατήματος που περιλαμβάνει την προφορία ότι όλοι οι εκπρόσωποι, ε, μάλλον όλοι οι ε, υπήκοοι της ε, χώρας αυτής έχουν το δικαίωμα στην απαλλαγή αυτή. Και μετά, αν μείνει αυτό, τότε μπορεί να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετική πράξη με την οποία η χώρα μπορεί να μεταφερθεί στο παράθυμα που περιλαμβάνει τον κατάλογο των χωρών εκείνων που δεν ε, έχουν απαλλαγή από προξενική θεώρηση. Το θέμα ποιο είναι. Όπως εξηγήσατε εσείς με μεγάλη ακρίβεια, το ζήτημα ήταν ότι αυτό το ενδιάμεσο βήμα της αναστολής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι αυτό είχε την ε, μορφή ε, εφαρμοστικής πράξης και δεν θα έπρεπε να γίνει λοιπόν με κάτι πράξη. Και θεώρησε ότι η χρήση αυτής της τεχνικής για να τροποποιηθεί το παράρτημα ήταν τεχνικό μέσον για να φτάσει τελικά στη χρήση κατεδουσιοδότησης πράξεων. Το δικαστήριο απέριψε την προσφυγή και έχουμε κάπως περισσότερες πληροφορίες τώρα για, δίνει μάλλον περισσότερες πληροφορίες για τον διαχωρισμό μεταξύ κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων Γνωρίζετε ότι τώρα όλο αυτό το θέμα έχει καθυστερήσει και πολλές διαπραγματεύσεις και είναι και κάτι το οποίο εμφανίζεται ξανά και ξανά ως κόλλημα σε όλες τις νομοθετικές διαπραγματεύσεις. Όσο λοιπόν πιο ξεκάθαρες ενδείξεις έχουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τόσο καλύτερα έτσι ώστε να μπορείτε να στοχεύετε τις προσπάθειές σας στην ουσία των θεμάτων και να μην περνάτε τον χρόνο σας με το αν μια πράξη είναι εκτελεστική ή όχι. Το, η ιδέα ήταν αυτή η προοδευτική διαδικασία, δηλαδή προσωρινή, προσωρινός αποκλεισμός ορισμένων πολιτών να καταλήγει τελικά σε νομοθετική τροποποίηση. Αυτό που γνωρίζουμε τώρα, καλύτερα από πριν, ποιο είναι. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όσοι ήταν υποχρωμένοι να εγκρίνουν την κατευθυντική στην πράξη δεν είχε περιθώριο διακριτικό περιθώριο. Και αυτό σήμαινε στην ουσία ότι είναι εκτελεστική πράξη. Αυτό το απέρριψε το ε, δικαστήριο με τρόπο ξεκάθαρο και απρόσμενο. Χρησιμοποίησαμε μια φράση που δεν αναμέναμε εμεί. Είπε δηλαδή ότι ούτε η έκταση, ούτε η ύπαρξη του περιθωρίου διακρίσεως έχει είναι ουσιώδες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξεταστεί δηλαδή ως κριτήριο για μια πράξη αν είναι εκτελεστική ή ε, κάτι εξοδότηση. Νομίζουμε ότι αυτό είναι υπερβολικό διότι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία εάν ο βασικός κανονισμός δεν είναι ολοκληρωμένος τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξουσιοδότηση. Ανάμεσα λοιπόν σε ένα νομοθέτημα που δεν είναι ακόμα ε, ολοκληρωμένο μπορούμε να κατανοήσουμε ότι όπου ο κανονισμός δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένος, το περιθώριο εκείνων που καλούνται να τον εφαρμόσουν, να τον ολοκληρώσουν δηλαδή, μπορεί να είναι μεγαλύτερο. μεγαλύτερο. Και είχαμε την ευκαιρία επίσης να μέσω της αποφάσεως του δικαστηρίου να λάβουμε και κάποιες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό ή όχι. Το δικαστήριο λέει είτε προσωρινό είτε όχι, η φύση είναι ίδια για όλα εκείνα τα εκατομμύρια ανθρώπων στην τρίτη χώρα οι οποίοι θα δουν να αλλάζει η νομική τους κατάσταση, η αλλαγή αυτή εξισώνεται με το, εάν, με το ενδεχόμενο η χώρα τους να φύγει από το καλό παράτημα να πάει στο κακό παράτημα. Ακόμα και αν είναι προσωρινό. Αυτό λοιπόν είναι αρμοδιότητα του νομοθέτου να μεταφέρει την χώρα από το ένα παράτημα σε άλλο. Όσοι λοιπόν το πράττουν αυτό, τότε το πράττουν κατ' του νομοθέτη. Αυτό, ε, με αυτό το εξισώνει το δικαστήριο. Από την άλλη μεριά, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ότι το δικαστήριο θεωρεί ότι οι συνέπειες αυτής της αναστολής είναι ταυτόσιμες από κάθε άποψη, οδηγούν δηλαδή σαν η χώρα να μην απολάμβανε την απαλλαγή από την προξενική θεώρηση. Η τροποποίηση του βασικού κανονισμού, διότι περί αυτού επρόκειτο, το ερώτημα για μας είχε τελειώσει από την αρχή. Τώρα το δικαστήριο το ξαναλέει μετά από την υπόθεση Γιούρες ότι κανείς δεν μπορεί να τροποποιήσει το ε, περιεχόμενο του κανονισμού με ε, εκτελεστική πράξη. Εάν το αγγίξετε το περιεχόμενο του κανονισμού σημαίνει εξουσιοδότηση. Λέει η Επιτροπή, ναι, το αγγίξαμε το περιεχόμενο, αλλά τι κάναμε τελικά. Το δικαστήριο λέει είτε υποσημείωση ήταν αυτό που αλλάξατε είτε όχι, το γεγονός ότι η νομική κατάσταση των ε, ενδιαφέρων προσώπων αλλάζει είναι αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Αυτό θεωρεί λοιπόν ότι πρέπει να ξεκαθαρίζεται στο ίδιο το παράρτημα. Και άρα είναι κάτι εξουσιοδότηση στην πράξη. Πολλά από τα πράγματα αυτά φαίνονταν εξ αρχής προφανή. Τώρα, γιατί έχουν σημασία να ξαναλεχθούν στην απόφαση του δικαστηρίου, ότι δηλαδή κανείς δεν μπορεί να τροποποιήσει το περιεχόμενο ε, βασικού κανονισμού παρά μόνο κατ' εξουσιοδότηση. Διότι στις διαπραγματεύσεις βλέπετε καμιά φορά να εμφανίζονται επιχειρήματα ότι αν δηλαδή η τροποποίηση είναι ελαφράς μορφής δεν πειράζει, το κάνουμε και με εκτελεστική πράξη. Προφανώς λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Σημαντικό είναι επίσης διότι μπαίνει, μπαίνει επιτέλους ένα τέλος στον μύθο ότι είναι, υπάρχει ελευθερία επιλογής μεταξύ εκτελεστικής ή της πράξη. Το δικαστήριο λοιπόν καθαρά ότι δεν υπάρχει ελευθερία επιλογής. Ο νομοθέτης έχει ένα περιθώριο διακρίσεως, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 290 και 291. Όταν λοιπόν στους τριμερούς διαλόγους σας βλέπετε κάποιους συνομιλητές σας να λένε ότι «Αχ, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως είναι ε, ελευθερία επιλογής και γι' αυτό ζητούμε εκτελεστική πράξη», τώρα να είστε ακόμα πιο σίγουροι ότι δεν ισχύει αυτό. Ούτε μπορούσε άλλωστε ποτέ να είναι, ποτέ δεν υπήρξε, ποτέ δεν υπήρξε τέτοιο περιθώριο διακρίσεως δηλαδή και τώρα ξέρουμε ότι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι δεν θα είναι ποτέ περιθώριο διακρίσεως. Το περιθώριο διακρίσεως όπως είπαμε δεν είναι κριτήριο λοιπόν για να δει κανεί αν πρόκειται για εξουσιοδότηση ή όχι. Ο προσωρινό χαρακτήρα επίση δεν αλλάζει την φύση και, παραπάνω, και πάνω απ' όλα η διαμόρφωση του βασικού κανονισμού είναι μονάχα υπόθεση της νομοθετικής αρχής. Μπορούμε δηλαδή να συνοψίσουμε εν τέλει την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγοντας ότι ναι, πρόκειται για τροποποίηση, περιλάβατε ένα παράρτημα, μα ζητείτε να τροποποιήσουμε το παράρτημα, αλλά το ζήτημα αυτό πράγματι πρέπει να ενταχθεί σε παράρτημα. Πράγματι πρόκειται για τροποποίηση παρατήματος. Αν λοιπόν τώρα είχαν ικανοποιηθεί τους ισχυρισμούς τους αυτούς, ή της Κομισιόν δηλαδή, τότε θα ήταν πολύ ατυχές η νομοθετική αρχή δεν θα είχε το δικαίωμα ούτε καν να διαμορφώνει το περιεχόμενο του κανονισμού, να αποφασίζει αν θα περιληφθεί στον κανονισμό ή όχι, ή αν θα πρέπει αυτός να ενημερωθεί όχι, να επικαιροποιηθεί όχι. Επειδή όμως διαφυλάχθηκε εν τέλει το δικαίωμα αυτό, ότι το, η νομοθετική αρχή μονάχα διαμορφώνει το περιεχόμενο του κανονισμού, αυτή τη στιγμή κάποιο αγγίξει τον κανονισμό, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πράξη κατεξουσιοδότηση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα κάνατε για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν κανένας συνάδελφος θέλει να λάβει τον λόγο επ' αυτού, όχι. Μήπως η Κομισιόν, η Κομισιόν, η Κομισιόν. Τότε ευχαριστώ τις κοινοβουλευτικές υπηρεσίες για την παρουσίασή τους. Πριν τα διάφορα θα ήθελα να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, το έκανα ήδη τρεις φορές, αλλά ξανά. Αλλά και στο προσωπικό και σε όλους τους άλλους. Και στους ερμηνευτάς. Τους ευχαριστώ και αυτούς για τη σκληρή τους εργασία. Καλά Χριστούγεννα λοιπόν. εκ μέρους της σκληρότερα εργαζομένης επιτροπής του Κτηνοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Τα διάφορα τίποτα. Δευτέρα 11 Ιανουαρίου η πρώτη μας συνεδρίαση στις 15 η ώρα.